Diamo inizio allora. Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ. Καλώς ήρθατε, αγαπητά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητά επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πραγματικά είμαι πολύ ευτυχής που σας υποδέχομαι για αυτή την διακοινοβουλευτική συζήτηση για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι εδώ παρόν και ο ε, Πολωνός Υπουργός Γεωργίας Μάρεξ τον οποίο τον ευχαριστώ και τον καλωσορίζω. Η μεταρρύθμιση την οποία προετοιμάζουμε είναι η πρώτη στα 50 χρόνια της ιστορίας της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής, την οποία οι βουλευτές διαδραματίζουν ένα τόσο σημαντικό ρόλο. Όπως γνωρίζετε, η Συνθήκη της Λισαβόνας κατέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνομοθέτη στο τομέα της γεωργίας σε ίσο επίπεδο με το Συμβούλιο, αλλά επίσης ε, ενίσχυε σημαντικά το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, ιδίως μέσω του νέου μηχανισμού ελέγχου της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 12 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χαίρομαι παρατηρώ ότι οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια χρησιμοποιούν ενεργά αυτά τα νέα δικαιώματα. Η γεωργία είναι ο τομέας όπου τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν παρουσιάσει το μεγαλύτερο μέρο διολογημένων γνωμοδοτήσεων και άλλες συνεισφορές. Ελπίζω ότι η σημερινή συζήτηση θα μας οδηγήσει στο να κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς τα μπρος στην κοινή μας προσπάθεια για να ξεύρουμε απαντήσεις στις νέες προκλήσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπίσει σήμερα το νέο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Πώς ε, να αντιμετωπίσουμε την ε, επιστηστική ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, τη βιοβικιλότητα και τα άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα και την αναγκαιότητα να διατηρήσουμε μια εδαφική ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ε, να πρασινίσουμε τις ενισχύσει της ΚΑΠ, ε, να τις καταστήσουμε πιο νόμιμες και πιο ισότιμες ε, και δικές στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών, πώς να προσαρμόσουμε τα εργαλεία της αγοράς για να αντιμετωπίσουμε την μεγάλη διακύμανση των τιμών των αγροτικών προϊόντων και πώς να διασφαλίσουμε την επιβίωση των αγροτικών κοινοτήτων ε, στην Ευρώπη στα πλαίσια ενός παγκοσμίου ανταγωνισμού. Πιθανότατα όλοι θα γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με την έκθεση Αλμπερντές στις 23 Ιουνίου την ε, θέση του για την ε, κοινή αγροτική προτιμητική προς το 2020, μέχρι το 2020. Αυτή η έκθεση που υποστηρίχθηκε από ευρία πλειοψηφία στην Ολομέλεια είναι η επίσημη απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Νοεμβρίου του 2010. Και επίση συνάδει με προηγούμενη θέση για το μέλλον τη ΚΑΠ μετά το 2013 που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2010. Έκθεση του κυρίου Λάιον. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα στοιχεία κλειδιά της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πολύ συνθετικό τρόπο. Συμφωνούμε με τους στόχους της Κομισιόν για μια κοινή αγροτική πολιτική πιο πράσινη, πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα για μια μεταρρύθμιση της ΚΑΠ σύμφωνα με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Γεωργία και που να απαντά στα αιτήματα των πολιτών ε, για να λάβει μια νέα νομιμότητα. Συμφωνούμε συνολικά με την προσέγγιση που προτείνεται από την Κομισιόν στην ανακοινωσή της. Υπό το φως των μελλοντικών προκλήσεων χρειαζόμαστε μια ισχυρή και βιώσιμη κοινή αγροτική πολιτική και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατάλληλη, επαρκής ε, χρηματοοικονομική πόρη, έκθεση DES όπως και έκθεση ΛΑΙΟΝ και πιο πρόσφατα η έκθεση Γκαρίγα της Επιτροπής Σούρα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο υπογράμμισαν ε, ότι ο προϋπολογισμός, ε, γεωργικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διατεθεί στο ίδιο επίπεδο όπως το προϋπολογισμός του 2013. Και αυτή είναι η επιθυμία μας. Δηλαδή να μπορέσουμε να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο αυτό η ανησυχία που εκφράσαμε χθε μάλιστα στον Επίτροπο Ντέτσεν Τσόλο για την πρόταση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που παρουσίασε η Κομισιόν στι 29 Ιουνίου. Γιατί αυτό το πάγωμα ε, δεν αποτελεί κατά τη γνώμη μας ένα πραγματικό πάγωμα των πόρων, αλλά περικοπή ε, των πόρων για την κοινή γεωργική πολιτική σε πραγματικούς όρους. Έτσι λοιπόν δεν ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά η πρόταση της Κομισιόν ε, πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο αφετηρίας για διαπραγμάτευση. Εμείς ε, θα προσπαθήσουμε να την τροποποιήσουμε προκειμένου να έχουμε τους απαραίτητους πόρους για μια μεταρρυθμίση που θα μπορεί να εγγυθεί την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων, την ε, αηφορία της γεωργικής παραγωγής και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των γεωργών και των καταναλωτών στην Ευρώπη. Αγαπητοί συμμετέχοντες, αγαπητά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. συμπρασματικά θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία μας ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ε, αναφέρεται στην έκθεσή μας, οι συνεισφορές που έχουν στελεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια, μπορείτε να τα βρείτε στο φακελό σας και η σημερινή συζήτηση θα ε, είναι χρήσιμα στοιχεία για να βοηθήσουν την Κομισιόν στο να προετοιμάσει τις νομοθετικές της προτάσεις που θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο. Εν τέλει, πριν να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Γερουσίας, της, Πολωνικής Γερουσίας, τον κύριο Τζέρτζε Γέρζη Κροσινόφσκι, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες σημαντικές πληροφορίες για το πώς θα ζητάτε το λόγο. Έτσι, έτσι όλοι όσοι έχουν εγγραφεί Ακόμη και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρουν ε, πέρα από το φάκελο ε, που έχουν δύο κάρτες για να ζητήσουν το λόγο. Η πράσινη κάρτα είναι για το πρώτο γύρο και η κόκκινη κάρτα για το δεύτερο γύρο της συζήτησης. Καλό όλους όσους θέλουν να πάρουν το λόγο να ε, γεμίσουν μία από αυτές τις κάρτες και να τη δώσουν το συντομότερο δυνατό στους κλητήρες. Όπως ε, μπορείτε να δείτε έχουμε πάνω από 50 ε, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν εγγραφεί και θα μπορούσαμε ίσως ε, να μην, ε, δεν θα μπορούσαμε ίσως να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα. Πάντως θα βάλουμε τα δυνατά μας για να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον ένα αίτημα λόγου ανά Εθνικό Κοινοβούλιο να καλύπτεται. Για να τα καταστήσουμε όλα αυτά δυνατά θα ήθελα να σας ζητήσω σε όσους πάρετε το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτηση, να μην υπερβείτε το χρόνο ομιλίας σας. Δηλαδή πρέπει να περιοριστείτε στα δύο λεπτά. Λοιπόν, θα σα ε, δώσω κάποιε περαιτέρω ενδείξεις όταν θα έχουμε λάβει όλα τα αιτήματα του λόγου και φυσικά θα βλέπετε και το χρόνο που θα τρέχει στην οθόνη. Σα ευχαριστώ όλου, σα ευχαριστώ για την πολύ μεγάλη συμμετοχή, για την αθρά συμμετοχή. Α ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτησή μα και με επαναλάβω, θα ήθελα να δώσω το λόγο κατευθείαν στον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας ε, της Γερουσίας της Πολωνίας, τον κύριο Γέρσκι Κροσκικόφσκι. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές ε, και Βουλευτές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση και ξέρετε πως ε, μόλις αναλάβαμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής ε, η συζήτηση για το μέλλον της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 κατέδειξε πω υπάρχει ανάγκη να έχουμε μια ισχυρή πολιτική η οποία θα μπορέσει να εγγυηθεί την ανάπτυξη και όχι τη στασιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί αυτή η πολιτική, θα πρέπει να είναι δίκαιη, ισόνομη και να εγγυάται ίσως όρου ανταγωνισμού μεταξύ των αγροτών όλων των κρατών μελών. Κυρίες και κύριοι, στις συζητήσεις οι οποίες συνεχίζονται για την κοινή γεωργική πολιτική δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ε, η πολιτική αυτή δεν είναι μόνο για τους αγρότες αλλά και για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφασίζουμε να έχουμε μια πολιτική η οποία θα είναι πιο κατανοητή από όλους και θα παρουσιάζει πιο ξεκάθαρα τα Οφέλη που προσφέρουν οι αγρότες στην κοινωνία, γιατί οι αγρότες δεν έχουν μόνο ευθύνη για την παροχή τροφίμων, αλλά και για το περιβάλλον, για την προστασία του τοπίου, των ζώων και της βιοποικιλότητας. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναμένουν ε, και έχουν βεβαίως προσδοκίες η γεωργία να παράγει ασφαλή προϊόντα υψηλούς ε, ποιότητες. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει η ευκαιρία όχι μόνο στις ε, μεγάλες εκμεταλλεύσεις αλλά και στις μικρές εκμεταλλεύσεις να μπορέσουν να βελτιστοποιήσουν την ε, παραγωγή τους. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι μεταρρυθμίσεις να μην είναι μόνο μικρές αλλαγές αλλά να είναι σημαντικές και ουσιαστικές βελτιώσεις για συγκεκριμένους ε, κλάδους οι οποίοι συχνά είναι περιθωριοποιημένοι οι δημοσιονομικές προοπτικές που έχουμε παρουσιάσει από το 2013 έως το 2020 βλέπουμε πως έχουν μία μείωση κατά 10% των ε, κονδυλίων της ε, σύγκλησης και από ό,τι φαίνεται δεν ε, πάμε προς μια πλήρη εξίσωση των άμεσων πληρωμών, κάτι το οποίο είναι ανισχυτικό δεν θα πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των ε, κρατών μελών και θα πρέπει να υπάρχει τελικά μια ισότητα πληρωμές σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαφοροποίηση βάσει ιστορικών ε, κριτηρίων και βεβαίως ε, δεν συμφωνεί με την ε, αρχή της ε, αλληλεγγύης ούτε με τις αρχές του ανταγωνισμού εάν μιλάμε για μια ενιαία αγορά. Στον πρώτο πυλώνα δε της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι σημαντικό να δούμε το τι γίνεται για ε, την ε, κατανομή αυτών των άμεσων πληρωμών μεταξύ των ε, κρατών μελών και να δούμε βέβαια και την δυνατότητα να εφαρμοστεί το ίδιο σύστημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή των πληρωμών μεταξύ των ε, κρατών μελών. Θα πρέπει να φύγουμε από τα τωρινά κριτήρια που αφορούν ε, ιστορικές ποσότητες παραγωγής και να περάσουμε σε ένα σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων με βάση τους ε, τωρινούς στόχους της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Στην δε συζήτηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή είχαμε τους ε, πολίτες Ένωσης οι οποίοι τονίζουν τον ρόλο που θα πρέπει να έχουν οι άμεσες πληρωμές μετά το 2013. Η εφαρμογή περιβαλλοντικών στόχων, το λεγόμενο πρασίνισμα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πρέπει όμως να σημειώσουμε πως ήδη τώρα λαμβάνουν οι αγρότες ε, άμεσες πληρωμές για την εφαρμογή περιβαλλοντικών στόχων στόχων μέσω της λεγόμενης πολλαπλής συμμόρφωσης. Και θα πρέπει να σημειώσουμε την συνεισφορά των ε, μικρών ε, εκμεταλλεύσεων. Η δε σύνδεση των πληρωμών με τους περιβαλλοντικούς στόχους δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο να έχουμε δυσανάλογα βάρη τα οποία θα επιβληθούν ειδικά στις ε, μικρές εκμεταλλεύσεις. Θα πρέπει να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των περιοχών της υπαίθρου και της γεωργίας, κάτι το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να επιτύχουμε τους ε, στόχους της στρατηγικής του 2020. Θα πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε την εφαρμογή των ε, μέσων που υπάρχουν για τον εξυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των, ε, του τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων. και κύριοι, η Πολωνία, όπως ε, ξέρετε, ανέλαβε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι λοιπόν και οι προτεραιότητες μας για το δεύτερο εξάμενο του 2011 θα είναι η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, και στις άμεσες ε, πληρωμές και στον τομέα των στρεματικών ενισχύσεων. Και Βεβαίω ε, θα δούμε και τα τη κοινή αλληλευτική πολιτική Κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι εδώ πέρα ω πρόεδρο της Επιτροπή Γεωργία της Γερουσίας, Επιτροπή Γεωργία και Υπέθρου και είμαι επίσης ε, επικεφαλής ε, του Συνδικάτου Αλληλεγγύη που γιορτάζει φέτος τα 30 έτη του. Και ακούω κάθε μέρα τις απόψεις των ε, αγροτών. Οι αγρότες λοιπόν θέλουν να υπάρχουν ε, ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εξίσωσης των ε, άμεσων πληρωμών και της κατάργησης των μεταβατικών περιόδων. Οι αγρότες πιστεύουν πως οι μηχανισμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμή για τις απαιτήσει της πολλαπλής συμμόρφωσης επαρκούν για τους στόχους του πρασινίσματος, όπως το λέμε, και θεωρούμε θεωρούν πως ε, περαιτέρω απαιτήσει θα πρέπει να συνοδευτούν από περαιτέρω χρηματοδότηση. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πως χρειάζεται υψηλότερος προϋπολογισμός για την γεωργία και αναμένουν βεβαίως λιγότερα γραφειοκρατία και απλοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, αναμένουν επίσης μια φιλική και διάφανη πολιτική και διαδικασίας που θα είναι πιο κοντά στον αγρότη. Θεωρούν πως ε, θα είναι λογικό να υπάρξει μία εξορόψη για να μην υπάρχουν έντονες διακοιμάνσεις ε, τιμών στις αγορές. Αναμένουν ο ρόλος του αγρότη στην αλυσίδα ε, των τροφίμων να ενισχυθεί και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό. Κυρίε και κύριοι, θεωρώ πως θα πρέπει να ακούσουμε όλες αυτές τις φωνές και οι προσπάθειες ε, πολιτικών ε, και συνδικαλιστών θα πρέπει να συνδυαστούν για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση για να επιτύχουμε αυτές τις απαραίτητες αλλαγές. Τέλος, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω πως το Πολωνικό Κοινοβούλιο θα ήθελε βέβαια να συνεργαστεί με όλα τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε για την παρέμβασή σας ε, και τώρα να επενθυμίσω ότι σχετικά με το γλωσσικό καθεστώς είναι πλήρες το γλωσσικό καθεστώς. Έχετε δηλαδή ερμηνεία σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντεσαντζούλος που είναι αρμόδιος επίτροπο για τη Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ εφόσον υπάρχει δυνατότητα να εκφραστούμε σε όλες τις γλώσσες. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να συμμετέχω στην συνάντηση αυτή. Ακόμη και αν ε, πολλοί από εσά μιλούν εξ ονόματος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είχαμε ε, φυσικά ευκαιρία να συναντηθούμε και στις πρωτεύουσε ε, των ε, κρατών σας και φυσικά θα συνεχίσω να επισκέπτομαι τα κράτη-μέλη και να συναντώ και τους εκπροσωπούς των Εθνικών Κοινοβουλίων. Στο νέο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κοινή αγροτική πολιτική ενισχύεται ιδιαίτερα και ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να υπογραμμιστεί. Αυτή η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στις συζητήσεις δηλαδή και ε, στην προετοιμασία ε, για τη λήψη των μελλοντικών αποφάσεων. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι μια δημόσια πολιτική η οποία ενδιαφέρει το σύνολο του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι λογικό και χρήσιμο τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, να συμμετέχουν στη συζήτηση σε σχέση με αυτή την κοινοτική πολιτική. Ε, ίσως πρόκειται για την ε, μόνη ευρωπαϊκή πολιτική η οποία ασχολείται με ένα οικονομικό τομέα όπου οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν άμεσο αντίκτυπο στα κράτη-μέλη. Και έτσι λοιπόν καθίσταται ακόμη πιο σημαντική η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Έτσι λοιπόν, όπως γνωρίζετε, όταν ξεκίνησε η διαδικασία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε μια ευρεία συζήτηση, ίσως μια από τις ε, ευρύτερες συζητήσεις που έχει διοργανώσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ε, θίγησαν εκεί τρεις ε, στόχοι. Επισητιστική ασφάλεια, η ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την ποικιλομορφία των τροφίμων, ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσει η Γεωργία σε καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, γιατί εξορισμού η γεωργία, ξέρετε, λειτουργεί με φυσικούς σκοπόρους, βιοποικιλότητα, νερό, έδαφος και ο τρίτος στόχος για την ε, μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική είναι ο ρόλος που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την εξεύρυνση ισορροπίας ε, στην Ήπεθρο αυτούς τους προσανατολισμούς ε, θα τους βρείτε μεταφρασμένους, θα δείτε ότι συμπεριλαμβάνονται στην ε, ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα τέλη του περασμένου έτους και διαπιστώνω ότι αυτοί οι τρεις ε, στόχοι έχουν γίνει αποδεκτοί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα έγγραφα που έχουν υιοθετηθεί και εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή στην έκθεση του George Lyon όπως ε, και στην έκθεση του κυρίου Ντες. Και στις δύο αυτές εκθέσεις μπορούμε να δούμε τους ίδιους στόχους. Και καθίσταται όλο ένα και πιο σαφές ότι γύρω από τους στόχους ε, αυτούς οικοδομούνται οι προσδοκίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Βεβαίως, ε, παράλληλα με τις συζητήσεις για το περιεχόμενο της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους ε, για την επιτεύξη των στόχων αυτών. Από τη σκοπιά αυτή, το ότι η Επιτροπή δημοσίευσε τις δημοσιονομικές προοπτικές μέχρι το 2020, ή εκεί η κοινή αγροτική πολιτική είναι το κύριο σκέλος του προϋπολογισμού, η κυρία φωνή του προϋπολογισμού, δηλαδή διατηρείται ε, ότι είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για το 2013 με ένα περιθώριο σταθερότητας που προορίζεται σε άλλες δράσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πάντα για την ε, κοινή αγροτική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, όχι μόνο έλαβε υπόψη τις προσδοκίες ε, των κοινοβουλίων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών και των γεωργών σε σχέση με τη σημασία της παραγωγής τροφίμων και του ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίζει η γεωργία στην ευρωπαϊκή κοινωνία αλλά Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει μία από τις πλέον ε, συνεκτικές και συνεπείς ε, δημόσιες ε, κοινέ πολιτικές που προσδιορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο. Και έχουμε την ελπίδα ότι θα έχουμε κοινέ πολιτικές και για άλλες πολιτικές ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και συμφέροντος. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, προϋπολογισμό, εμείς ε, το φθινόπωρο θα παρουσιάσουμε και τις νομοθετικές προτάσεις ε, για την αναθεώρηση, για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Και στις προτάσεις αυτές θα συμπεριλαμβάνονται και οι λεπτομέρειες που θα αφορούν τους τρεις στόχους, ε, διατηρώντας φυσικά το ε, κύριο εργαλείο στήριξης των γεωργών, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις. Όμως ε, θα υπάρχει μια αναδιάρθρωση αυτών των άμεσων ενισχύσεων για να μπορούμε να απαντήσουμε πιο συγκεκριμένα στους στόχους της ΚΑΠ. Αυτές οι άμεσες ενισχύσεις, οι άμεσες πληρωμές που θα έπρεπε προσδιοριστούν, βάσει νέων κριτηρίων. Θα πρέπει να βάσει νέων κριτηρίων, δηλαδή δεν θα έχουμε πλέον τα κριτήρια της ε, παραδοσιακής παραγωγής, που δεν είναι πλέον κατάλληλα για τη σημερινή κατάσταση. Αυτά τα κριτήρια θα καθοριστούν με ένα τέτοιο τρόπο που οι γεωργοί να ενθαρρύνονται να επενδύουν στον τομέα της γεωργίας για να συνεισφέρουν ε, στην γεωργική παραγωγή για την οποία υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως ε, η γεωργική παραγωγή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους στόχους της ορθής διαχείρισης good management προκειμένου να πετύχουμε μία ανταγωνιστικότητα που θα περιλαμβάνει και οικολογικές πτυχές, όχι μόνο οικονομικές. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας μακροπρόθεσμα. Μαζί με τις ε, άμεσες ενισχύσεις που θα επαναπροσδιοριστούν, θα υπάρχει και ένα πιο προστευμένο σύστημα για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Ε, τώρα δεν ε, περιλαμβάνω εδώ τις εκμεταλλεύσεις που δεν παράγουν ε, για την αγορά. Εμείς θα προτείνουμε λοιπόν ένα απλουστευμένο σύστημα πληρωμών, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους γεωργούς, για να τους δοθεί κάποια ενθάρρυνση και κίνητρα να ασκούν μια σύγχρονη, μια μοντέρνα γεωργία. Μιλώντας ε, για το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Γεωργίας, πρέπει να σκεφτόμαστε φυσικά και το μέλλον ε, των αγροτών και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τους νέους επομένως. Πέρα από τις άμεσες ενισχύσεις ε, και τους μηχανισμούς της αγοράς, οι μηχανισμοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην καθημερινή κατάσταση της αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα στους γεωργούς ε, να ανταποκρίνονται στα μήνυματα της αγοράς. Θα πρέπει επίσης να αποκτήσουμε μέσα εργαλεία για την επιλύση των κρίσεων. Τελευταία διαπιστώσαμε ότι Αυτές οι κρίσεις ξεσπούν όλο ένα και συχνότερα και θα πρέπει να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο πακέτο, μια σύγχρονη δέσμη μέτρων ε, σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τις αγορές, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά σε περίπτωση κρίσεων και θα διατυπώσουμε νέες προτάσεις για νέα μέτρα. Πέρα από τη συνιστόσα αυτή, η γεωργική πολιτική έχει και μία ακόμη σημαντική συνιστόσα της ανάπτυξης της υπαίθρου, της αγροτικής ανάπτυξης για τον εξυγχρονισμό της γεωργίας. Το στοιχείο αυτό της ε, ΚΑΠ ε, θα είναι όλο ένα και πιο ενισχυμένο έτσι ώστε αφενός να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι στόχοι της στρατηγικής 2020 και αφετέρου να υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμών αρκετά ευρύ για τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορούν να πετύχουν τους στόχους αυτούς ε, σε περιφερειακό εθνικό επίπεδο. Για αυτό το δεύτερο πυλώνα θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προσδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επικλομορφία της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και σε ό,τι αφορά τις ε, δομές, τα είδη των ε, δομών, των εκμεταλλεύσεων των εταιρεών, όπως και τους διάφορους ε, παραγωγικούς τομείς. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη και στις περιφέρειες μέσω διαφορετικών μέτρων που θα βασίζονται στα μέτρα του δεύτερου πυλώνα να μπορούν να, να αναδιαρθρώσουν ε, τους γεωργικούς τομείς σε ορισμένες περιοχές ε, όπου ε, ο ρόλος των τομέων αυτών είναι σημαντικός από περιβαλλοντική σκοπιά. Και πριν να κλείσω θα ήθελα να επενθυμίσω ότι και στο μέλλον θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ενθάρρυνση θα πρέπει να ενισχύσουμε μάλλον περισσότερο το συνδέσμο μεταξύ της αγροτικής παραγωγής και της έρευνας και ανάπτυξης. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε την έννοια της γεωργίας της γνώσης, γιατί η αύξηση της αντιγνωστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, μια αηφόρος γεωργία, χρειάζεται και τη συνεισφορά της επιστημονικής έρευνας, ε, τη συνεισφοράς καινοτόμων ιδεών που θα είναι ικανές ε, να οδηγήσουν και σε νέες πρακτικές. Έτσι λοιπόν, ε, ο σύνδεσμος μεταξύ της εφαρμοσμένης έρευνας ε, και καινοτομίας και αγροτικών πρακτικών είναι κάτι που θα πρέπει να υποστηριχθεί μέσω χρηματοδότησης. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο προπολογισμό που προτείνεται προβλέπει για πρώτη φορά ένα αποθεματικό πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία. αλλά και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Θα υπάρχει λοιπόν συμμετοχή και των ερευνητών και θα υπάρχουν προγράμματα χρηματοδότησης 100%. Ε, ευρωπαϊκά προγράμματα που θα χρηματοδοτούνται 100% μέσα από όσα θα προτείνουμε από το σχέδιο της μεταρρύθμισης, ελπίζω να μπορέσουμε να ε, πετύχουμε τους στόχους που έχουμε καθορίσει. Όπως ε, από την αρχή της ε, θητείας μου, εγώ βασίζομαι πάρα πολύ στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί η μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να είναι πολύ πιο στοχευμένη από όσο σήμερα θα πρέπει να στοχεύει πολύ περισσότερο ε, και να ανταποκρίνεται στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και στις ελπίδες των Ευρωπαίων πολιτών. Αξίζεται πραγματικά το χειροκρότημά μας, ε, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε και για τη συνεχή βούλησή σας να διατηρείτε άμεση επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ ολοκληρώνεται ο πρώτος ε, γύρος των παρεμβάσεων δίνοντα το λόγο στον κύριο Αλμπερντέ, ο οποίος είναι ο εισηγητή τη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον ε, της ΚΑΠ 2020. Παρακαλώ, Άλμπερτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Παύλο, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνομιλητές, χαίρομαι ως ε, εισηγητής ε, του Ευρωπαϊκού Γενοβουλίου για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι το 2020 για το ότι βρήκαμε μία τόσο διακομματική ε, λύση. Γιατί βεβαίως Βλέποντας μεγάλες διαφορές στην Ευρώπη, αναρωτήθηκα πώς θα γίνει με αυτές τις μεγάλες διαφορές σε 27 κράτη-μέλη να μπορούσουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση που θα δεχτούν όλες οι ομάδες. Αλλά πρώτα απ' όλα στην Επιτροπή Γεωργίας είχαμε ευρεία συνένεση με 90% νομίζω των ψήφων για τις συμβαστικές λύσεις και ανάλογο ποστό και στην Ολομέλεια και νομίζω πως όλοι οι συνάδελφοι που εργάζονται στα κοινοβούλια μπορούν να αντιληφθούν πόσο δύσκολο είναι με τις διαφορές που υπάρχουν στην Ευρώπη να έχουμε τέτοιες πλειοψηφίες. Αλλά θέλαμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα για το μέλλον της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής και επίσης είχαμε τη θέληση να εκμεταλλευτούμε τη νέα κατάσταση μετά τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας και να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση η ξεκάθαρη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, ένα σαφές μήνυμα και η Κομισιόν και προς την Κομισιόν και θέλουμε να στηρίξουμε βέβαια τον Επίτροπο αλλά και προς το Συμβούλιο πως εδώ πέρα έχει αυτοπεποίθηση το Κοινοβούλιο και θα φανεί αυτό και τους επόμενους μήνες. Η έκθεσή μου βασίζεται στο ότι είναι αποστολή της Ευρωπαϊκής Γεωργικής Πολιτικής και αυτό το τονίζουν όλοι οι ομιλητές να εξασφαλίσει την διατροφική ασφάλεια για πάνω από ε, μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους. Επίσης, βάση αποτελούσε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει την πιο αηφόρο γεωργία σε ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να το ξέρουμε αυτό, αν και υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε ορισμένες τομείς. Πρέπει λοιπόν εκεί όπου υπάρχουν ε, ελλείψεις ε, να τις ε, καταπολεμήσουμε. Αλλά βάση της έκθεσης ήταν η γνώση πως μέχρι το 2050 παγκοσμίω θα πρέπει να ανεβεί η παραγωγή τροφίμων κατά 70% όπως μας λένε οι επιστήμονες. Και βάση αποτέλεσε επίσης πως στο παρελθόν η αύξηση της παραγωγικότητας ε, δεν έλαβε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε άλλα μέρη. Θα αναφέρω κάποια νούμερα από τον ΦΑΟ στη Ρώμη. Από το 1976 μέχρι το 2008 η, Ευρω... η παραγωγή δημητριακών στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1%. Στην Ασία κατά 97% ακόμη μεγαλύτερη διαφορά στην παραγωγή κρέατος. Στην Ευρώπη είχαμε μία αύξηση τα 32 αυτά χρόνια 6%. Στην Ασία 385% και αν τώρα θέλουμε να διαμορφώσουμε μια γεωργική πολιτική η οποία θα κάνει καψόνια στον Ευρωπαίο αγρότη για να παράγει λιγότερο τότε λέω πως ε, θα αποτύχουμε στην προστασία και των ζώων και του κλίματος και οποιοδήποτε άλλο πράγματος, γιατί πουθενά άλλου δεν τηρούνται αυτές οι προδιαγραφές όπως στην Ευρώπη. Αυτά ήταν η βάση ολόκληρης της έκθεσης. Έχουμε λοιπόν λάβει σημαντικές αποφάσεις κύριε Επίτροπε και ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας ε, στηρίξουμε. Το Κοινοβούλιο, όχι μόνο η Επιτροπή Γεωργίας που είναι φυσικό, ολόκληρο το Κοινοβούλιο ζήτησε να ε, διατηρηθεί το τωρινό ύψος στον μελλοντικό προϋπολογισμό της Γεωργίας. Τώρα, όπως φαίνονται τα πράγματα με την πρώτη αξιολόγηση των προτάσεων της Κομισιόν, φαίνεται πως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και βλέπω πως υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι ε, περικοπής. Ε, είχαμε και το Γερμανικό Συνέδριο των Αγροτών ε, και μιλήσει εκεί με την καγκελάριό μας και τώρα ε, βασιζόμαστε σε μια χρηματοδότηση του 1,05% ε, του ΑΕΠ και ε, έρχεται η Άγγελα Μέρκελ και μας λέει ανώτατο όριο πρέπει να είναι 1% του προϋπολογισμού. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην γίνει αυτό για να μην οδηγηθούμε σε περαιτέρω περικοπές στην γεωργική πολιτική ασφάλεια των τροφίμων λοιπόν είναι βασικός όχος της κοινή μας έκθεσης και εδώ πέρα θέλουμε να συνεισφέρουμε έτσι ώστε τα 500 εκατομμύρια καταναλωτές να μπορούν να βασίζονται στο ότι θα έχουν υγιή τρόφιμα τα οποία θα παράγονται με τρόπο αηφόρο. Άλλες αποστολές αναφέραμε ε, σήμερα το πρωί με τον Πολωνό Υπουργό τον κύριο Σαβίτσκι είναι η ενεργειακή αυτή αλλαγή που γίνεται και θα συμμετάσχει σε αυτήν και η γεωργία. Και αυτό σημαίνει μεγάλες προκλήσεις. Αυτό το οποίο τονίσαμε στην έκθεσή μας ε, και κύριε Επίτροπε οπωσδήποτε εδώ πέρα θα συμφωνείτε θέλουμε να διατηρήσουμε μια δομή δύο πυλώνων και στο μέλλον και νομίζω πως θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός αυτών των δύο πυλώνων η απλοποίηση αναφέρεται σε ολόκληρη την έκθεση. Θέλουμε ένα σύστημα άμεσων πληρωμών και στο δεύτερο πυλώνα που δεν θα οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία. Ως βουλευτής επί σειρά ετών γνωρίζω πως ε, δεν θα πρέπει καμιά φορά να τολμάμε να αναφέρουμε τη λέξη μείωση της γραφειοκρατίας στους αγρότες μας γιατί συμβαίνει συνεχώς το αντίθετο. Οπότε, αποστολή της Κομισιόν Κοινοβουλίου και Συμβουλίου είναι επιτέλους να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή τη γραφειοκρατία. Πρέπει να γίνει λιγότερη γραφειοκρατία και νομίζω πως έτσι μπορούμε να έχουμε μια πολύ σωστή προσέγγιση. Παραδείγματος χάρη φαντάζομαι πως ε, εάν είναι σημαντικό θέμα ο έλεγχος μπορούμε να λάβουμε μέτρα τα οποία ε, πιθανώς ε, θα βασίζονται στην πολλαπλή συμμόρφωση και εάν βγάλουμε αυτά τα μεγάλα θέματα νομίζω ε, μπορούμε να οδηγηθούμε σε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν χρειάζεται παντού πολλαπλή συμμόρφωση. Εάν απλώνουμε παντού αυτή την ε, πολλαπλή... Εάν, με συγχωρείτε, αφαιρέσουμε την πολλαπλή συμμόρφωση από την ε, εξάπλωση η οποία υπάρχει τελευταία, νομίζω υπάρχει χώρος για διαφορετικές ε, πολιτικές. Σημαντικό κομμάτι επίσης ε, των σκέψεών μας. Δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένα νούμερα όσον αφορά τις διαφορές των άμεσων ε, πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών. Κοιτάξτε όμως, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν τόσες, ε, τόσο μεγάλες διαφορές, να πάμε από τα 100 στα 500 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή ε, η ψαλίδα μεταξύ των ε, κρατών μελών. Πρέπει να κλείσει αυτή η ψαλίδα χωρίς μεγάλες μεταβατικές περιόδους, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα για να έχουμε περισσότερη δικαιοσύνη. Αλλά αυτό το οποίο με εξέπληξε είναι πως ε, δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μόνο μεταξύ κρατών μελών στις άμεσες πληρωμές, αλλά μου προξένησε εντύπωση το ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές εντός των κρατών μελών στις άμεσες πληρωμές. Εάν ε, πάρουμε ως παράδειγμα την Ιταλία. Είναι κάποιοι στη Βόρεια Ιταλία, στο Νότιο Τυρόλο, πληρώνονται 50 ε, ευρώ το εκτάριο και στην ε, Λομαρδία 500-600. 500-600 δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αν ε, παραμείνει έτσι η κατάσταση και κάποιοι πληρώνονται π.χ. για την καλλιέργεια δημητριακών 500-600 ευρώ και κάποιοι άλλοι 100-200 ε, το συμπέρασμα είναι σαφές ε, και να σας πω και κάτι άλλο από γερμανική σκοπιά εμείς αποφασίσαμε στη Γερμανία πως μέχρι το 2013 από τις ε, αρωτρές περιοχές θα πάνε στις υπόλοιπες περιοχές 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και το αποδέχτηκαν οι αγρότες, δεν υπάρχει μεγάλη συζήτηση και αυτό οδηγεί και σε μεγαλύτερη ισότητα εντός ε, του, των κρατών μελών. Επίσης ζητήθηκε η απομάκρυση από τα ιστορικά και μεμονωμένα σημεία αναφοράς. Στην έκθεση επίσης ε, αποφασίσαμε την αναγνώριση των μικρών αγροτών και του ρόλου που παίζουν. Και εδώ πέρα βλέπουμε κύριε Επίτροπε πως δεν καταφέρατε παρόλη την θέληση να βρείτε έναν κανονισμό για το τι είναι μικρός αγρότης σε 27 χώρες. Η κατάσταση στη Λετωνία είναι τελείως διαφορετική από την Ελλάδα ε, βλέποντας και την πρώην συνάδελφο εδώ πέρα αυτό το οποίο θεωρείται μικρός αγρότης στην ε, Λετωνία μπορεί να είναι μεγάλη εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λέμε πως θα πρέπει σε ε, εθνικό επίπεδο να ορίζεται ποιος είναι ο μικρός αγρότης. Όσον αφορά δε τον έλεγχο αυτών για το πρασίνισμα. Και πάλι εδώ πέρα βλέπετε ότι δεν μπορούμε να ισχύουν τα ίδια πράγματα στην Σικελία και τη Φιλανδία. Είναι πιο διαφορετικές δεν γίνονται. Δηλαδή αν απογειωθεί κανείς με το αεροπλάνο από το Ελσίνκι, σκέφτηκα κύριε Επίτροπε τι άλλο πρασίνισμα θέλουν να κάνουν οι Φιλανδοί. Όλη η χώρα είναι πράσινη. Όταν απογειώνεται κανείς από την Κατάνια σκέφτηκα τι γράφουμε, τι λέμε 30% πρασίνισμα στους ε, Πρώτα απ' όλα πρέπει να φέρουμε νερό στο νησί πριν μιλήσουμε για πρασίνισμα. Ε, τίποτα άλλο δεν μπορώ να φανταστώ. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορές στην Ευρώπη αν είναι να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Μία παρατήρηση επίσης για τις αγορές. Εμείς δώσαμε ιδιαίτερα μεγάλο βάρος στην διατήρηση των μέσων της ε, αγοράς. Αυτό δεν το λέω τώρα επειδή το είπαμε διακομματικά. Χρειαζόμαστε πράγματι αυτά τα μέτρα παρέμβαση στην αγορά, ειδικά για περιπτώσεις ε, κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτείτε γιατί η ε, οικονομική αντιμετώπιση η οποία υπάρχει στην Κομισιόν είναι σωστή, αλλά από πλευράς όγκων δεν επαρκεί για να μπορέσει να υπάρξει μια σωστή παρέμβαση στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα κονδύλια εδώ πέρα. Επίσης, στις ε, συζητήσεις ζητήσαμε ο Οργανισμός Οργάνωσης ε, Αγοράς Ζάχαρης να παρατηθεί μέχρι το 2015 και να ε, ξανασυζητήσουμε τα φυτοαιγειονομικά. Επίσης αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους G20 λέμε πως χρειαζόμαστε παγκόσμιες λύσεις για να εμποδιστεί η τεράστια κερδοσκοπία με τα τρόφιμα και τις γεωργικές πρωτοσύλλες. Εντάξει, κερδοσκοπία υπάρχει πάντα, αλλά όταν μιλάμε για κερδοσκοπία η οποία γίνεται στις ε, χρηματαγορές πρέπει να εμποδιστεί για να μην γίνεται εις βάρος των τροφίμων. Επίσης, η ανάπτυξη της υπαίθρου, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να εξασθενήσει ο δεύτερος πυλώνας, πρέπει αντιθέτως να ενισχυθεί γιατί είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και εδώ πέρα βέβαια πρέπει να ληφθούν υπόψη διαφορές μεταξύ χωρών και περιφερειών. Επίσης ζητήσαμε οι μειονεκτικές περιοχές να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται μέσω του δεύτερου πυλώνα. Κύριε Μπέντροπε, κύριε Τσιόλος, αναμένουμε λοιπόν τώρα τις νομοθετικές σας ε, προτάσεις, θα τις παρακολουθήσουμε ως κοινοβούλιο και θα ήθελα να κλείσω με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Υπουργό το πρωί και που το λέω και εγώ και μου ασκούν Κοιτάξτε, εάν, βλέπουμε τις, εάν δούμε τις διαφορές ε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, απέχουμε πάρα πολύ από μια κοινή γεωργική πολιτική. Ελπίζω να επιτύχει λοιπόν η μεταρρύθμιση για να γίνει πράγματι κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. E Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τώρα να ξεκινήσουμε τις παρεμβάσεις ε, των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο σε τρία μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και σε ένα συνάδελφο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Άννα ε, πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης ε, από, την, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασίλειου. Παρακαλώ. Good afternoon, Chairman. Χαίρετε σε όλους. Ε, βρίσκω ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία σε όλες τις εκθέσεις, ε, κυρίως εκθέσεις του Κοινοβουλίου που έχουν υποβληθεί εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης. Ε, σε σχέση με αυτά που μας είπε ο εισηγητής ο κύριο Ντές, θα έλεγα το εξή. Μα μίλησε για τη ρύθμιση και για την κατάργηση τη πολλαπλή ε, συμμόρφωση ουσιαστικά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να εξετάσουμε και δεν έχει εξεταστεί ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να στηρίξουν του νέου αγρότε ε, και τη νέα γενιά αγροτών. Επίσης, έκκληση προς απλούστευση απευθύνατε Νομίζω έτσι θα νομιμοποιηθεί περαιτέρω το σύστημα και το θέμα ότι υπάρχει ε, ομοθυμία σε σχέση με την ανάγκη της επισητιστικής ασφάλειας και της στρατηγικής σημασίας που έχουν τα τρόφιμα ε, θα αποτελέσουν τον πυρήνα της συζήτησής μας ε, και αυτή είναι η βασικότερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το αναφέρουμε στην έκθεσή μας σχετικά με την πράσινοποίηση σε εισαγωγικά θα πρέπει όλοι να υποφεληθούν από την αλλαγή δηλαδή να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, αλλά ταυτόχρονα να αυξηθεί και η βιωσιμότητα, ενώ ταυτόχρονα απλουστεύουμε και αφαιρούμε ε, τα διοικητικά, τα γραφειοκρατικά άχθη, ούτως ώστε να έχουμε πραγματικά αγροπεριβαλλοντικά ωφέλη και όχι ε, αυξημένη πολλαπλή συμμόρφωση μπορούμε να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλήξουμε σε αποφάσεις που θα είναι υποφελείς ε, και για τους πολίτες ε, και για τον κόσμο της Γεωργίας και για τους καταναλωτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αν Μαϊκίντος. Ε, πολύ, πολύ σεβαστήκατε και το χρόνο σας ε, μέχρι τελευταίου λεπτού. Τώρα θα ακούσουμε από το Ιταλικό Κοινοβούλιο τον κύριο Πάολο Ρούσο. Μικρόφωνο παρακαλούμε για τον ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ΚΑΠ ε, δεν ε, θα πρέπει ε, απλώς ε, να χρησιμοποιεί ότι δίνουμε απλώς εισόδημα σε μια κατηγορία Ευρωπαίων πολιτών. Ε, η εκταμείευση των απαραίτητων πόρων είναι απαραίτητη για μια Ευρώπη που δεν είναι ικανή να παράγει τρόφιμα και τροφή σε συνδίκες απόλυτης εχνασιμότητας και ασφάλειας και επίσης σε ευξανόμενους ρυθμούς και ε, επίσης χρειάζεται και μια πολιτική προσέγγιση που θα ευνοεί ε, την ανάπτυξη της υπαίθρου ως μοντέλο ανάπτυξης ε, και εκεί θα διασφαλίζουμε και την ιστορία και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μια απαραίτητη απέτηση που να προτείνει έναν ηθικό τρόπο ανάπτυξης. Πρέπει να εκπαιδευτούν περισσότεροι πόροι για να καλυφθούν οι απαιτήσει των σημερινών αγροτών Όπω των Ιταλών εργοντών. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε εδώ το εξή ότι αν ε, ε ότι το θέμα της ε, έρευνα και της ανάπτυξη, αν δεν ληφθούν αυτά υπόψη, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, θα έχουμε ένα σύστημα αποστοδρομικό. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο και καινοτόμο σύστημα. Ταυτόχρονα πρέπει να ξανασκεφτούμε ε, το θέμα θέμα ε, ενός ε, ε, μη επαγγελματικού κλάδου, δηλαδή να μην λαμβάνουν τις ίδιες ενισχύσεις ε, συνεχώς ε, οι ίδιοι άνθρωποι που δεν παράγουν. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε για το όφελος των καταναλωτών, ε, να ουσιαστικά και να προσδώσουμε περισσότερη αξία στους τόπους και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε Ρούσο. Δίνω τώρα το λόγο στον Πρόεδρο ε, της Επιτροπής Γεωργικών Υποθέσεων από το Λιθωνικό Κοινοβούλιο, τον κύριο Πούπνης. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ε, ευχαριστούμε για αυτή την ε, συνάντηση, ειδικά τον κύριο Ντεκάστρο. Εάν δούμε την κοινή γεωργική πολιτική, τότε τα μέτρα του πρασινίσματος θα δείτε πως είναι πάρα πολύ φιλόδοξα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια σε ένα κοινό πλαίσιο, αλλά η ανάγκη για ποιοτικά τρόφιμα υπάρχει και αυτή, οπότε οι στόχοι του πρασινίσματος ε, και τα ποιοτικά τρόφιμα είναι εξίσου σημαντική στόχη. Τώρα το κομμάτι του πρασινίσματος στις άμεσες ε, πληρωμές δεν νομίζω ότι αποτελεί ιδιαίτερα ετοιμολογημένη βάση γιατί ε, νομίζω πως ε, μπορεί να επηρεάσουν έτσι ολόκληρη τη χρηματοδότηση ειδικά σε χώρες ε, που δεν έχουν ακόμα ανανεώσει επαρκώς την παραγωγική τους βάση. Οι άμεσες ε, πληρωμές ε, θα πρέπει νομίζω να, να αποτελέσουν στόχο προτεραιότητας στην κοινή πολιτική και μία δίκαιη μέθοδο για την κατανομή που θα πρέπει να βρεθεί για να μην έχουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού γιατί τα παλαιά κράτη-μέλη εξακολουθούν να προτιμώνται και βεβαίως να έχουν μειονέκτημα τα νέα κράτη-μέλη. Οπότε έχουμε μεγάλες ανησυχίες λόγω αυτής της ε, ε, περίοδου μέχρι το 2020 που θα χρειαστεί για να εξωθούν οι πληρωμές. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η περίοδος. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Και τώρα είναι η σειρά των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή τη επιτροπή. Ο κύριο Χόσλινγκ ε, θα πάρει το λόγο που είναι επικεφαλή τη ομάδα των Πρασίνων στην επιτροπή αυτή. Παρακαλώ, Μάρτιν. <laughs> Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα ε, μπορώ να σου πω, η κοινή γεωργική πολιτική είναι πλέον ε, υπό έλεγχο εφόσον έχει συναπόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ότι έχουμε ευρύτατη βάση για το σχέδιο αυτό έκθεση σημαίνει πως είμαστε πολύ φιλόδοξοι και νομίζω υπόθηκε ήδη στην έκθεση πως θα πρέπει να γίνει πιο πράσινη και πιο δίκαιη η κυνηγερική πολιτική. Βεβαίως έχουμε το θέμα της κατανομής το οποίο θα μας απασχολήσει στις ε, συζητήσεις ε, που έρχονται και στα κράτη-μέλη και στην Γεωργία γιατί βεβαίως έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αδικίες που πρέπει να αναφερθούν. Βεβαίως ε, μιλήσαμε για κάποιο πλαφών, αλλά βρήκαμε νομίζω μία λύση για να διατηρηθούν και στις μεγάλες επιχειρήσεις θέσεις εργασίας και να υπάρχουν και καλύτερες περιβαλλοντικές επιθώσεις. Αυτή είναι η βάση των συζητήσεων που έχουμε και προς τα εκεί ελπίζω να πάμε. Τώρα ε, αναφέρθηκε ήδη το πρασίνισμα κατά 30% είναι μια τάξη μεγέθους που νομίζουμε μπορεί να υπομειστεί η Ευρωπαϊκή Γεωργία και ελπίζω να συνεισφέρει η γεωργία και στρατηγική βιοπικιλότητας και την προστασία του κλίματος, πράγματα τα οποία δεν πρέπει να παραμελήσουμε και σημαντικά γιατί δικαιολογούν την γεωργία για την χρηματοδότηση της γεωργίας στην κοινή γνώμη. Θα ήθελα όμως να αναφέρω κάτι, να το συζητήσουμε ανοιχτά. Νομίζω πως μπορούμε να συζητήσουμε το ότι θα πρέπει η Γεωργία να αυξήσει την παραγωγή της κατά 70% τη στιγμή που 15% των τροφίμων πετυχαίνεται. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη για αηφόρο Γεωργία και θα πρέπει να υπάρξει μια έρευνα σε αυτόν τον ε, τομέα, να υπάρξει μια πολιτική έρευνα, ειδικά προς την κατεύθυνση της αηφορίας. Ευχαριστώ. Μάλιστα, θα επιστρέψουμε στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η κυρία Μπατζελή έχει το λόγο, είναι και συνάδελφος, ε, πρώην συνάδελφος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τώρα εκπροσωπεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχηθώ ε, κουράγιο και καλή δύναμη στον Προεδρεύοντα της, ε, του Συμβουλίου, όπου έχουν μια πολύ σκληρή εργασία μπροστά τους και στον κύριο Ντές, ο οποίος ε, πραγματικά παρουσίασε μια σημαντικότατη έκθεση, όπου αξιώνει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία συναπόφασης με τα άλλα θεσμικά όργανα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι κανένας από εμάς δεν θεωρεί ότι η κοινή αγροτική πολιτική το 2014 και 2020 θα είναι η ίδια αγροτική πολιτική όπως ήταν τα τελευταία δέκα χρόνια. Περνάμε σε μια Ευρώπη όπου έχουμε ένα νέο μοντέλο οικονομικής και θεσμικής διακυβέρνησης, χρηματοδότησης του κοινοτικού προπολογισμού με διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετικό τρόπο κατανομής των πόρων στα κράτη-μέλη, όπου πλέον σε αυτή τη νέα χρηματοδότηση του κοινοτικού προπολογισμού εμπλέκεται ή εύχομαι να εμπλακεί και το χρηματοπιστωτικό σύστημα με τη φορολόγηση του, ε, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα ήθελα να θέσω ορισμένες αρχές τις οποίες θεωρώ ότι ως Εθνικό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα το προτάσουμε αλλά και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το διαπίστωσα και στην έκθεση του κύριου Ντές. Ποια είναι η αγωνία των αγροτών. Εάν θα μπορούν να βγουν πλέον στις αγορές. Η στήριξη καθαρά και μόνο από τον κοινοτικό προπολογισμό δεν είναι πρωταρχικό μέλημα πλέον του Ευρωπαίου αγρότη, ακόμα και του Έλληνα αγρότη. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ο στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ο έλεγχος της αγοράς της διατροφικής αλυσίδας. Ποιοι όμως θα διαχειριστούν αυτό το σύστημα. Και στην έκθεση του κύριου Ντες αναφέρεται ο προσδιορισμός του ενεργού αγρότη του ενεργού πολίτη, αυτός ο οποίος δεν διαχειρίζεται μόνο περιβαντολογικά τη γη, αλλά παράγει αγροτικά διατροφικά προϊόντα. Και στο βαθμό που έχουμε διατροφικά προϊόντα πρόκειται περί μιας μεγάλης ανταγωνιστικότητας και μιας μεγάλου αγώνα εντός του τοπίου. Δεύτερο, για το κόστος της παραγωγής. Κριτήριο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση των αγροτών πετρέλαιο, ενέργεια αυξάνεται, συνεπώς θα πρέπει να εγκριθούν και φορολογικές απαλλαγές. Και κλείνω με το εξής για το δεύτερο πυλώνα. Θεωρούμε ότι πρέπει να τελειώσει ο τρόπος της πασπερμίας των μέτρων στο δεύτερο πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης και να υπάρχει δυνατότητα ολοκληρωμένων διαρθρωτικών προγραμμάτων τα οποία θα συντάσει ο κάθε, η κάθε περιφέρεια και η κάθε εθνική αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Μπετζελή. Τώρα το λόγο έχει εκπρόσωπο τη Γερουσία Τσεκή Δημοκρατία, Αντωνίου Μασταλήρ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση της ε, σημερινής συνάντησης που έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη γνώμη μου διότι θα ε, πρέπει στο μέλλον να ενισχύσουμε τις ε, σχέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ώψη της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα να σας εκθέσω εν συντομία τη θέση της τσεχικής γερουσίας για αυτό το θέμα. Η γερουσία μας εδώ και καιρό ασχολείται με το ζήτημα Έχουμε μελετήσει διάφορα ευρωπαϊκά έγγραφα σε συνδυασμό με την κυβέρνηση και με τους εκπροσώπους των ενώσεων των γεωργών και νομίζω ότι συμφωνούμε επί των στόχων που έχουν προσδιορίσει το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, τα προσεχή χρόνια χρειαζόμαστε μία βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, μια βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και ε, οφείλουμε επίσης να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και να επιδείχουμε μια ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη στην ε, Ήπεθρο. Αυτά συνάδουν με την στρατηγική Ευρώπη 2020 και εξάλλου αυτή είναι η θέση και της τσεχικής κυβέρνησης. Θεωρούμε ότι οι δαπάνες θα πρέπει να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και νομίζουμε ότι η κατανομή των δαπανών θα πρέπει να είναι 80 και 20% αντίστοιχα για τον πρώτο και για τον δεύτερο πυλώνα. Προτείνουμε λοιπόν το 80% να διοχετήσουμε στοχεύονται στου αγρότε και το 20% στο δεύτερο πυλώνα στην πρασινοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής στην ανάπτυξη τη υπαίθρου. Δηλαδή, επίσης η έννοια της προθέσπιση ανωτά του ορίου, το περίφημο κάπινγκ σε σχέση με το μέγεθος μιας γεωργικής ε, εκμετάλλευσης, ε, θα λέγαμε το εξής ε, 77 εκτάρια είναι η μεγαλύτερη γεωργική εκμετάλλευση στην Τσεχία που είναι και μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο προσδιορισμό του ανωτάτου ορίου θα πλήξει με τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις ε, στη χώρα μας. Ε, δεν μπορεί η Γερουσία ω εκ τούτου να προσυπογράψει αυτή την πρόταση για τη θέσπιση ανωτάτου αερίου. Για τον πρώτο πυλώνα δε συμφωνούμε με τη συγχρηματοδότηση και για τα πρώτα χρόνια μετά το 2013 κυρίω, διότι Ε, θα πρέπει να προβλέψουμε και μια μεταβατική περίοδο, ώστε να μην ε, ε, υποστεί κανένα κράτο μέρο διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τι άμεσε πληρωμέ. Την κρίση μα θα πρέπει να τη βασίζουμε σε αντικειμενικά κριτήρια και σε θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ερβέ Γκεμάχαντ που εκπροσωπεί ε, το, το Γαλλικό Εθνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Τσιόλος, τον κύριο Ντέσε για τη στρατηγική θεώρηση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Εγώ θα τη συνοψίσω σε τέσσερις λέξεις, στα γαλλικά βέβαια. Φιλοδοξία πρώτον, σε σχέση με τους στόχους της κατοχύρωσης επιστημιστική ασφάλειας, δημοσιονομική φιλοδοξία για να έχουμε επαρκή πόρους στη διάθεσή μας και να αποφύγουμε τις απόπειρες επανεθνικοποίησης της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, και τέλος ε, αποφυγή διπλών πληρωμών στις ε, πολυμερείς, είτε πρόκειται για τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις είτε για τις διμερείς διεθνείς διαπραγματεύσεις, διότι η Ένωση έχει σημειώσει Μεγάλη πρόοδο στον τομέα του εμπορίου ε, σε παγκόσμια κλίμακα. Ε, Δεύτερο πυλώνα, ανάπτυξη τη υπαίθρου. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι διατηρεί τη ισορροπία ανάμεσα στου δύο αυτού πυλώνε και συμμεριζόμαστε το στόχο τη ε, πρασινοποίηση των στόχων του πρώτου πυλώνα, στο μέτρο που θα είναι απλά τα μέτρα, αρμονικά και θα εφαρμόζονται παντού σε όλη την επικράτεια τη Ένωση με ομοιόμορφο τρόπο. Τρίτη προτεραιότητα, η ρύθμιση, η κανονιστική ρύθμιση που δεν πρέπει να περιορίζεται συγγνώμη, σε ένα μινιμαλιστικό δίχτυ ασφαλείας. Το αντίθετο πρέπει να είναι ε, καινοτόμα ε, ούτω ώστε να είναι πιο, ε, πιο ευέλικτα τα εργαλεία της αγοράς, να αντιδρούμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να χειριζόμαστε καλύτερα τη ζήτηση καθώς και την δημόσια και ιδιωτική αποθεματοποίηση. Ε, Κλείνοντα θα ήθελα να κάνω κάποιες πολύ ειδικέ παρατηρήσεις. Πρώτον για την εκτινοτροφία. Η εκτινοτροφία στη Γυρία Ήπειρο μπορεί να περιέλθει σε ακόμη δυσχερέστερη θέση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να διατηρηθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσει. Θα θέλαμε επίσης στον πρώτο πυλώνα να υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσεις για τις ε, ε, μειονεκτούσες περιοχές, κυρίως για τις ορεινές περιοχές. Θα θέλαμε επίσης ο ε, τομέας να προστατευτεί με διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης ε, και τέλος για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες θα επιθυμούσαμε να ληφθούν όντω υπόψη οι ιδιαιτερότητές του Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα είναι σειρά προσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χέρμπερτ Ντόρφμαν. Sí, grazie signor Presidente. Ja, ich denke, das ist ja eine sehr interessante Phase, die wir derzeit. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον στάδιο σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να αναφέρω δύο θέματα. Κάτι που ήδη αναφέρθηκε από τον Αλμπερτέ η κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των δύο πυλώνων θα πρέπει να παραμείνει εντός των κρατών μελών. Όμως εδώ στην Επιτροπή μας εμείς ε, μιλήσαμε κυρίως για την κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως μεταξύ των παλιών και των νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως στην πραγματικότητα ε, πραγματικά ε, τα κράτη-μέλη δεν έχουν προβεί σε κατάλληλη κατανομή των κονδυλίων στο ιστορικό τους και πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό γιατί είναι γεγονό ότι πολλά κράτη-μέλη κυρίω όσα κράτη-μέλη είναι σε καλύτερη κατάσταση είναι αυτά που λαμβάνουν περισσότερους πόρους για να ικανοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Πρέπει να το φροντίσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Τώρα από την άλλη είχαμε μια ιδιαίτερα φιλελεύθερη πολιτική τελευταία και αυτό μας οδήγησε οι ποσοστώσεις στο γάλα, στη ζάχαρη και λοιποί μηχανισμοί είτε να περιοριστούν είτε να εξαλειφθούν η δική μας επιτροπή και ήταν και παρόν και πρόεδρος, έστειλε μια αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τόσο χάρη στο γαλακτοκομικό τομέα στι Πολιτείες, ε, σχεδιάζεται μια ρύθμιση γιατί δεν λειτουργεί ε, ο ενώ Εμείς χάσαμε αυτά τα συστήματα στη δική μα Ήπειρο, δηλαδή θα πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτό το τόσο φιλελεύθερο χαρακτήρα τη κοινή ε, γεωργικής πολιτική. Εγώ νομίζω ότι το να πετάξουμε από το παράθυρο όλα αυτά τα συστήματα που έχουν δείξει τη χρησιμότητά τους τελευταίες δεκαετίες δεν είναι το πλέον λογικό. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Ντόρφμαν και τώρα θα επιστρέψουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρτ Λίντεν που εκπροσωπεί το Γερμανικό Κοινοβούλιο, τη Γερμανική Κατουβουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφώς τάσσονται υπέρ μιας κρατεάς κοινή γεωργικής πολιτικής στο μέλλον. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος και του Γερμανικού Κοινοβουλίου για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τα κονδύλια στο τωρινό τους επίπεδο στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να απλουστεύσουμε την κοινή γεωργική πολιτική γιατί ε, συνιστά ένα μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος ε, για τα κράτη-μέλη. Ως προς τις άμεσες πληρωμές ε, με δικαιούχους στα κράτη-μέλη, προσοχή διότι στην ε, Γερμανία οι άμεσες πληρωμές αντιστοιχούν στο 60% ε, ε, των αμέσων ενισχύσεων και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια διαρκή στήριξη του εισοδήματο των γεωργών. Όμως σε μεγάλο βαθμό είναι αποσυνδεδεμένα τα εισοδήματα των γεωργών από την παραγωγή και σε αυτό προστίθενται τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα για αυτό το λόγο θα πρέπει να ε, επιλέξουμε τα μέτρα ε, πρασινοποίησης ε, με ιδιαίτερη προσοχή και να εξασφαλίσουμε μια ευρή υποστήριξη για την κοινή γεωργική πολιτική από τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πάση θυσία πρέπει να αποφύγουμε την αύξηση της γραφειοκρατίας και με τον εξορθολογισμό και την απλούστευση κοινή γεωρικής πολιτικής θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στη Γερμανία. Έχουμε ήδη κάνει ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις ε, ε, ομοιόμορφες ενισχύσει των ε, γεωργών. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την προστασία της φύσης και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 πρέπει να συνδυαστεί με την κοινή γεωργική πολιτική για να έχουμε μια βιώσιμη γεωργία η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες ε, της αγοράς. Γι' αυτό οι επιχειρήσεις βάση ενός νέου κανονισμού, οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να πλήττονται από τη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Τώρα εκ μέρου του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, Γκέρτ Κάουμπερτ, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ε, συζήτηση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, είναι πάρα πολύ σημαντική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για τις ε, αγροτικές περιοχές της Ευρώπης ε, και για το εισόδημα των αγροτών μας. Πολλά πρέπει να έχουμε κατά νου. Πώς παίρνει το σχάρι το θέμα της ε, άνησης κατανομής του κέρδους κατά μήκος της αλυσίδας. Το Κοινοβούλιο επικεντρώθηκε στην προστασία των καταναλωτών, ασχολήθηκε με την προστασία των καταναλωτών, όμως ε, πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά. Οι συνάδελφοι από την Κομισιόν και το Κοινοβουλίο πρέπει να εργαστούν για να υπάρχει πιο ισορροπημένη νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Αυτό που θέλουμε τελικά είναι ευημερία και στην υπεθρό έτσι λοιπόν ε, πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές ε, στην πολιτική ανταγωνισμού και αυτό θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με τη μεταρρύθμιση της κάψας. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο του κοινοβουλίου, στην εκπρόσωπο του Συνοβουλίου της Σουηδίας, την κυρία Μπρόντεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μα δίνετε να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα και ευχαριστώ για όλε αυτέ τι ε, πολύ ενδιαφέρουσε ε, παρεμβάσει. Έχετε αναφερθεί ήδη ε, στα μεγάλα ζητήματα, ανάπτυξη τη υπαίθου, επιστημιστική ασφάλεια, προστασία των πολιτών και των γεωργών. Θα τα καταφέρουμε μεταρρυθμίζοντα την κοινή γεωργική πολιτική να συνδυάσουμε όλα τα ζητούμενα, δηλαδή ανάπτυξη τη υπαίθου, προστασία του περιβάλλοντο και προώθηση της γεωργίας. Ακούσαμε ήδη κάποιες απαντήσεις. Οι γεωργοί θα πρέπει να συμβάλλουν. Ναι, συμφωνούμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολλά, ε, πολύ μεγάλες οι προκλήσεις, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία της βιοπικιλότητας ε, και όταν μιλάμε για το δεύτερο πυλώνα, ανάπτυξη της υπαίθρου, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ανάπτυξη, η έρευνα και η γεωργία είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν κατά προτεραιότητα στο μέλλον ε, και πρέπει να αναδειχθούν σε προτεραιότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορεί να συμβάλλει ούτως ώστε να έχουμε μια βιώσιμη γεωργική παραγωγή ε, και στις τρίτες χώρες, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ισχύσουν ομοιόμορφα κριτηρία σε όλα ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθηθούν και τα ε, ίσα δικαιώματα των γυναικών σε σχέση με τους άντρες. Νομίζω ότι θα χρειαστεί δημοσιονομική στήριξη από πλευράς όλων μας για να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει το εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλτη Τζιγμάντα. Δεν είναι από την Επιτροπή αυτή, έτσι, λοιπόν, από την Επιτροπή αυτή. Ζητώ συγγνώμη για την προφορά του ονόματό σα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στον κόσμο της πολιτικής και χαίρομαι πάρα πολύ που συζητούμε για τους γεωργού χωρίς να ξεχνάμε την ανταγωνιστικότητα. Ανοίξαμε τις ε, αγορές μας. Ε, όταν μπήκαμε στην, Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε πλέον και επιτρέψαμε την απελευθέρωση του τομείς, όχι όμως ε, στη Γεωργία, στη Λιθουανία. Η Γεωργία εγκατέλειψαν τη γεωργία και πέρασαν σε άλλους παραγωγικούς τομείς. Έτσι λοιπόν έχουμε 100.000 λιγότερους απασχολούμενους ε, στον τομέα της γεωργίας. Όσοι ήταν ε, στο παρελθόν γεωργοί τώρα εργάζονται παραδείγματος χάρη σε σερβιτόροι, σε εστιατόρια. Και εγώ πιστεύω λοιπόν ε, ότι είναι πολύ θετικό να υπάρχει μια μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και Πιστεύω ότι η Πολωνική Προεδρία θα πετύχει τους στόχους της και θα είναι πιο δίκαιη στο μέλλον ε, η μεταρρύθμιση της ΚΑΠΗ. Οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να κατανεμώνται με πιο δίκαιο τρόπο. Πρέπει να εγγυηθούμε τις ε, θέσεις εργασίας. Ε, οι γεωργοί θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους, με το λειτουργήμά τους και θα πρέπει να παράγουν τον πλούτο που χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε και για να πετύχουμε μια επιστηταστική ασφάλεια και μια ασφάλεια στον εφοδιασμό των τροφίμων, γιατί πολλές φορές αγοράζουμε τρόφιμα από το εξωτερικό χωρίς να γνωρίζουμε την ποιότητά τους. Πρέπει να ανοίξουμε την κυνηγερική μας πολιτική, όμως ε, διατηρώντας την απαραίτητη ρύθμιση, έτσι ώστε η ΚΑΠ ε, να συνεχίσει να αποτελεί πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας. Μάλιστα, τώρα θα δώσω το λόγο και πάλι στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ισμαντ Βιέστιους Λιέγκης, από τη Λετωνία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να λάβουμε και εμείς ε, μέλος στην συζήτηση αυτή. Το ΔΕ Κοινοβούλιο μας και η κυβέρνηση χαιρετίζει την ανακοίνωση του Επιτρόπου Τσόλους και ζητούμε μια μεταρρύθμιση του συστήματος άμεσων πληρωμών για να είναι δίκαιο και να μην βασίζεται πλέον σε ιστορικά κριτήρια έτσι ώστε οι μεγάλες ανισότητες στη στρεματική ενίσχυση να μειωθούν. Έχουμε τώρα την ανακοίνωση της Κομισιόν για το πολιετές μουσιονομικό πλαίσιο για την Ευρώπη του 2020 ως βάση περαιτέρω συζητήσεων. Δυστυχώς, οι τελευταίες αυτές προτάσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές έχουν ως κίνδυνο να χαθεί η ευκαιρία το να γίνει το σύστημα άμεσων πληρωμών πιο ανταγωνιστικό και δίκαιο. Γιατί οι διαφορές ε, μεταξύ πληρωμών ε, ε, των κρατών μελών εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε η σύγκληση θα πρέπει να είναι και τολμηρότερη και ταχύτερη ξεκινώντας από το 2014. Δεν έχει φτάσει ο καιρός να καταργηθεί η αδικία ε, τη στιγμή που οι πλούσιοι αγρότες στη Δυτική Ευρώπη πληρώνονται πολύ περισσότερο από τους αγρότες στη Βαλτική και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συνάδελφοι. υπό το φως των ε, πιθανών επιπτώσεων για τους λετονούς αγρότες ε, των προτάσεων της Κομισιόν, η... το κοινοβούλιο μας, το οποίο κανονικά έχει διακόψει για το καλοκαίρι, θα συνεδριάσει εκτάκτως αυτή την Πέμπτη. Θα εκφράσουμε τη σοβαρή μας ανησυχία για τις ε, τελευταίες προτάσεις της Κομισιόν, οι οποίες θα χρειαστούν πάρα πολύ ρύθμιση για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες οικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, ειδικά μεταξύ των αγροτών μας. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα από το Βουλγαρικό Εθνικό Κοινοβούλιο η κυρία Κριστίνα Ιβάνοβα Γιάντσεβα. Παρακαλώ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής για τη χώρα μας. Είμαι σχετικά νέο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να επιμείνουμε. Οφείλουμε να υφετήσουμε μια ομοιόμορφη προσέγγιση για το σύστημα των άμεσων πληρωμών ούτω ώστε να τύχουν ισότιμη μεταχείριση, δίκαιη μεταχείριση όλοι οι γεωργοί. Οι πληρωμέ ε, για την ε, Βουλγαρία θεωρούμε ότι θα πρέπει να φτάσουν στο ανώτατο όριο το 2014 και όχι το 2016. Αυτό δεν αποτελεί βάρος ε, για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και αντίθετα θα στείλει ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα προς τους γεωργούς μας, ε, οι οποίοι θα συνειδητοποιήσουν ότι την χάνουν δίκης μεταχείριση σε σχέση με τους γεωργούς άλλων χωρών. Ως προς την πρασινοποίηση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής σίγουρα θα είναι χρήσιμη, αλλά θα πρέπει η πάση θυσία να αποφύγουμε την επικάλυψη με τον ε, δεύτερο πυλώνα. Ως προς την ε, χρηματοδότηση θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη στήριξη για να καλυφθούν ε, οι αυξημένες άμεσες πληρωμές οι ενισχύσει όμω ε, θα πρέπει να έχουν ω δικαιούχου μόνο του ενεργού γεωργού. Αφήστε που θα πρέπει να διευκρινίσουμε, να ε, ε, δημιουργήσουμε ένα σαφέστερο ορισμό για τον ενεργό γεωργό. Τι εστί ενεργός γεωργός. Επίσης, αυξημένη στήριξη προς τους μικρούς κλήρους. Ένα κάτι άλλο που ζητάμε και θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα κοινό ταμείο για την χρηματοδότηση αυτών των ενισχύσεων, αλλά αυτό θα πρέπει να ε, εκφεύγει των κονδυλίων ε, του τακτικού προπολογισμού τη Ένσου. Μάλιστα. Και τώρα εκπρόσωπο από το Εθνικό Κοινοβούλιο τη Μάλτα ε, θα πάρει το λόγο ο κύριο Φιλίπ Μίτσου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για τα νέα κριτήρια, για τις ε, ενισχύσεις, για τις πληρωμές. Νομίζω ότι τα κίνητρα για τους νέους αγρότες ε, και επίσης ε, η έρευνα και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία σύμφωνα με τις ε, απόψεις της χώρας μου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ισορροπημένη η ΚΑΠ. Θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία σε σχέση με τη σημερινή. Τα παλιότερα κράτη-μέλη και τα σχετικά νέα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρίσκονται θα πρέπει μεταξύ αυτών να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε τις ε, μεγάλες αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των ε, μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων και των μικρότερων. Οι τελευταίοι γεωργοί των μικρών εκμεταλλεύσεων πολλές φορές ε, δεν έχουν καν τα μέσα για για να εξασκήσουν το επαγγελμά τους. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος. Τώρα, τρίτο σχόλιο. Το τρίτο σχόλιο μου αφορά Ορισμένε ε, σκέψει μπορεί να έχουν ε, τα κράτη-μέλη στο ότι ένα μέγεθο ταιριάζει σε όλου. Στη Μάλτα όλε οι εκμεταλλεύσει, ε, όλε οι εταιρείε είναι μικρέ και όλοι οι γεωργοί δραστηριοποιούνται σε ευάλωτε, σε μειονεκτικέ περιοχές, Όμω θα πρέπει να ανταγωνιστούν με γεωργού από την Ευρώπη και από την Αφρική προέρχονται από μεγαλύτερε εκμεταλλεύσει. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να λάβετε υπόψη και την κατάσταση των μικρότερων κρατών μελών. Στη δική μας περίπτωση είναι τόσο μικρές εκμεταλλεύσεις που διακινδυνεύουμε με εξάλληψη της γεωργίας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Μάλιστα, ευχαριστώ και ας περάσουμε στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, αν έχετε το λόγο. Η Βουλή των Λόρδων στην έκθεσή της ήθελε να μιλήσει για την έρευνα, αλλά δεν έχει πολύ νόημα να επιδοτούμε την έρευνα εάν δεν πρόκειται να υιοθετηθεί. Και τι εννοώ, σταματάει η υιοθέτησή της από τους πράσινους ακτιβιστές, ε, καθώς ε, μιλάνε για Φραγκενστάιν και Τζίνι που θα βγουν από το μπουκάλι και τέτοια. Πρέπει να υπάρξει, να υψώσουμε λίγο ανάστημα και αν δεν γίνει αυτό η Βρετανική και η Ευρωπαϊκή Γεωργία θα μείνουν πίσω. Υπάρχει ακόμα η ψευδέστηση πώς ε, μπορούν ε, να επηρεάσουν και να ζεστάνουν τον παγκόσμιο καιρό οι αγρότες μέσω των εκπομπών ε, μεθανίου. Ανισχώ πάρα πολύ για αυτές τις ρυθμίσεις καθώς φαίνεται πως δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία αν δούμε τους τελευταίους πάρα πολύ κρύους χειμώνες παρά την αύξηση του διοξιδίου του ανθρακά. Αν δεν το παρασέξατε εσείς, εγώ έχασα το 1 τρίτο της οδιάς μου γιατί είχε παγώσει το έδαφος από το χιόνι. Τώρα, για την ε, τελευταία απαγόρευση την οποία έγινε για τα ε, για τα αυγά. Ε, αν υπάρχει κάνα άλλο τέτοιο παράδειγμα για το ότι τουλάχιστον εμείς ακολουθούμε τους κανόνες ενώ όλοι οι υπόλοιποι να μην πω τη χειρονομία κάνουν προς την ε, Κομισιόν δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην σας άρεσαν αυτά που είπα αλλά γλιτώστε το χρόνο. Μάλιστα, δώσατε το καλό παράδειγμα. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν, θα ακολουθήσουν οι βουλευτές από την Φιλανδία. Τον λόγο έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Δασών, Γιάρη Λέπα. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική εισαγωγική παρουσίαση που κάνατε. Στο μέλλον θα χρειαστούμε μια αποτελεσματική κοινή γεωργική πολιτική και γι' αυτό χρειάζεται παρκή σε χρηματοδότηση. Θα πρέπει να πληρούνται οι όροι βάσει των οποίων θα λειτουργήσει εξίσου το σύστημα σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κυρίως στις μειονεκτούσες ε, λόγω εδαφομορφολογικών συνθήκων ε, περιοχές. Στην Φιλανδία έχουμε πολύ περιορισμένες δυνατότητες ε, εκμετάλλευσης του εδάφους ε, και γι' αυτό έχουμε τις ε, ενισχύσεις που βασίζονται στον τρόπο παραγωγής και προορίζονται σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου δύσκολα μπορεί να καλλιεργηθεί το έδαφος. Αυτές οι ενισχύσεις ε, θα πρέπει εν μέρη να χρηματοδοτούνται από το δεύτερο πυλώνα και θεωρούμε ότι το ανώτατο όριο των 250 ε, ευρώ ε, θα πρέπει να είναι υψηλότερο Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε αντικειμενικά κριτήρια ως προς τον τρόπο υπολογισμού αυτών των ενισχύσεων. Τώρα, σε σχέση με τα πράσινα ε, στοιχεία της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής, ε, θα πρέπει να προσέξουμε για να μην επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά και άλλο τους γεωργούς, γιατί θα έχουμε περισσότερους γραφειοκράτες από ό,τι γεωργούς στο τέλος. Μιλήσαμε επίσης για την εξισορρόπηση των αναγκών της κοινή γεωργικής πολιτικής και των αναγκών των αγορών. Ε, σε σχέση με την καλλιέργεια του εδάφους ε, θα πρέπει να ισχύσουν και την παραγωγή ε, τροφίμων και την κτηνοτροφία θα πρέπει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τρίτες χώρες να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και χρειαζόμαστε γι' αυτό ένα κοινοτικό σήμα αλλά όχι μόνο για τα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης αλλά και τα προϊόντα των τρίτων χωρών. Σας ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στη Γερμανία και πάλι και θα δώσω το λόγο στην Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας ε, Τροφίμων και Καταναλωτών ε, του ε, Γερμανικού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, νομίζω όλες οι ομάδες στην Γερμανική Βουλή, ε, υποστηρίζουν ε, επί της αρχής την ε, πρόταση του κυρίου Ντες. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε πως η κοινή γεωρική πολιτική συνολικά ήταν πολύ επιτυχής για την ευρωπαϊκή κοινότητα και ειδικά για τη Γερμανία. Έχουμε αγροτική οικονομία υψηλών επιδόσεων σε όλα τα κρατήδια, εξάγουμε και παράγουμε με ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστασίας των ζώων και η παραγωγή είναι σε μεγάλο βαθμό αϊφόρος. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για διάθεση αγροτικών κονδυλίων αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Γνωρίζετε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επικριτική διάθεση, αλλά παρόλα αυτά ε, πράγματι πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη δικαιοσύνη, δεν είναι δυνατόν σε χώρες οι οποίες είναι ασθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά από τη Γερμανία να είναι τόσο μεγάλη η διαφορά στην ε, στρεματική ενίσχυση. Αλλά θεωρούμε πως ε, το μέσο το οποίο προτείνεται του πλαφόν δεν είναι το σωστό. γιατί αυτό το οποίο θα γίνει ότι θα καταλήξουν οι αγρότες να γίνουν λογιστές. Επίσης η σύνδεση με τις θέσεις εργασίας δεν νομίζω επίσης ότι στέκει. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι περισσότερη ειδική και όχι απλά εργατικά χέρια τα οποία θα απασχοληθούν κάπου. Το πρόβλημα του πρασινίσματος δεν παίζει μεγάλο ρόλο στην Γερμανία, ούτως ή άλλως 5% των εκτάσεων δεν επιτρέπεται να καλλιεργηθεί. Έχουμε πάρα πολλές μεγάλες ε, εκτάσεις σε αγρανάπαυση και ε, προστατευμένες εκτάσεις. Ε, οπότε θα πρέπει να δούμε το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε στις περιπτώσεις κρίσης επίσης για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια βοήθεια αν αυτή χρειάζεται. Σας ευχαριστώ. Και τώρα είναι η σειρά του Λουξεμβούργου, από το Εθνικό Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου. Θα δώσω το λόγο σε ε, κάποιο άτομο που γνωρίζουμε όλοι εδώ και χρόνια, στον κύριο Φερνάν Μποντέν, ο οποίος ε, είναι Υπουργός ή ήταν Υπουργός Ευχαριστώ. Παόλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για, γιατί διοργανώνει αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντέση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη που εξέφρασε εξ ονόματο ε, του Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική αναμφίβολα και ε, ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και επαρκή χρηματοδότηση. Οι δημοσιονομικές δε προοπτικέ όπως μα τις εκθέτει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστούν μια καλή βάση για τι μελλοντικέ διαπραγματεύσει στον τομέα αυτό και υποστηρίζουμε αυτή την προτεραιότητα ε, της επιστημιστικής ασφάλειας, ε, της ε, παραγωγής ποιοτικών τροφίμων, της βιώσιμης παραγωγής ποιοτικών τροφίμων είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μας, ε, να ακολουθήσει αυτήν την οδοευρωπαϊκή γεωργία της ταχύτητας, της αποτελεσματικότητας, της υλοποίησης των στόχων ε, της στρατηγικής 2020, ε, που θα συνδυαστεί με την νέα κοινή γεωργική πολιτική. Για την ίση κατανομή τώρα των άμεσων ενισχύσεων που είναι ένα απαραίτητο κομμάτι, ένα αναπόσπαστο τμήμα του εισοδήματος ε, των ε, γεωργών. Λοιπόν θα πρέπει αυτές οι ενισχύσεις να διοχετεύονται στους ενεργούς γεωργούς ε, για να έχουμε μία βιώσιμη αποτελεσματική πολιτική που σέβεται το περιβάλλον και προστατεύει τους φυσικούς πόρους θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα ο δεύτερο πυλώνα για τι άμεσε ενισχύσεις. Ε, έχουμε κάποια προβλήματα για αυτή τη σχέση του 30% των άμεσων ε, πληρωμών με τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που υπερβαίνουν τις τωρινές προϋποθέσεις. Εμά, στη χώρα μα, στο Λουξεμβούργο, έχουμε πάρα πολλά αγροπεριβαλλοντικά μέτρα στο δεύτερο πυλώνα και σχεδόν ε, όλοι οι γεωργοί συμμετέχουν σε αυτέ τι πρακτικέ, Εάν τώρα ένα τμήμα αυτών των αγροπεριβαλλοντικών κανόνων ενταχθεί στον πρώτο πυλώνα, δίχως όμω να αυξηθούν οι άμεσε ενισχύσει, αυτό συνεπάγεται απώλεια της τάξης σχεδόν του 30% του εισοδήματος των γεωργών, διότι δεν θα είναι πλέον δικαιούχοι των ενισχύσεων στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα και άρα θα πρέπει να βρούμε μία λύση διότι έχουν κάνει σοβαρότατες προσπάθειες αυτοί οι άνθρωποι στα πλαίσια του δευτέρου πυλώνα. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να ε, πληγούν η Γεωργία από τη μεταφορά των ενισχύσεων αυτών στον πρώτο πυλώνα το κομμάτι των πληρωμών που αντιστοιχεί στις μειονεκτούσες περιοχές τώρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα αντισταθμιστικών ενισχύσεων για τους γεωργούς μας, για τις μειονεκτούσες περιοχές. Εάν αυτό το τμήμα ενταχθεί στον πρώτο πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, δίχως όμως να αυξηθεί το όριο των άμεσων ε, πληρωμών και αυτό θα πλήξει το εισόδημα των γεωργών. Άρα θα πρέπει να βρούμε μια λύση, μια ένα περιθώριο ε, ελιγμών, ούτω ώστε τα μέτρα να κατανεμηθούν με καλύτερο τρόπο ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο πλάνο. Σα ευχαριστούμε, Φερνό. Θα μα περάσουμε τώρα στο Αυστριακό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή Γεωργία, Μάρτιν Πρένεντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και για την διοργάνωση αυτή τη συνεδρίαση που μα δίνει την ευκαιρία να τοποθετηθούμε. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το οποίο ήδη αναφέρθηκε για την διατήρηση δηλαδή των εξωτικών πληρωμών στο υφιστάμενο επίπεδο και νομίζω πως είναι σημαντικό αυτό όπως επίσης και θα πρέπει να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους καταναλωτές πως ε, το να έχουν ε, υγιή και ασφαλή τρόφιμα είναι ε, κάτι το οποίο πρέπει να πληρωθεί με μια τιμή που αντικατοπτρίζει το κόστος της παραγωγής. Πράγματι για το όλες που αναφέρθηκε χρειάζεται περισσότερη δικαιοσύνη αλλά υπάρχουν βεβαίως και διαφορετικά επίπεδα μισθών και κόστους ζωής στην κάθε χώρα και επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και βεβαίως διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες και μειονεκτήματα της ε, παραγωγής. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στην αγορά έτσι ώστε οι γεωργοί να μπορέσουν ε, να αντισταθμίσουν τις διακοιμάνσεις των τιμών με κάποια αποθήκευση καθώς ε, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να υπάρχει μια σταθερότητα τιμών για να μπορέσουν και αυτοί να επενδύσουν μακροπρόθεσμα για να υπάρχουν και προπτικές για τους νέους αγρότες και για τους καταναλωτές βεβαίως να υπάρχει και μια ασφάλεια όσον αφορά την προμήθεια των τροφίμων. Όσον αφορά δε το πρασίνισμα θα συμφωνήσω κάπως με τον ε, Λουξεμβούργιο συνάδελφο. Είναι ήδη αρκετά πράσινο το τοπίο στην ε, Αυστρία. Τα δε, τοπία των, τα δε ζήτημα των, του πρασινίσματος θα μπορούσαν να επεκταθούν νομίζω σε ολόκληρη την Ευρώπη και παραπέρα. Ξέρετε, παραδείγματο χάρη, πως και από πλευράς ε, μπορεί να αποφεληθεί ε, εδώ πέρα η χώρα. Σε διεθνές επίπεδο έχουμε ανοίξει ε, πάρα πολύ και νομίζω θα έπρεπε να ξαναδούμε πώς θα γίνει εθνική και περιφερειακή η γεωργία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Και τώρα επανέρθουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε από την Βουλή των Λόρδων στον Λόρδο Κάρτερ, πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας Ελίας και Περιβάλλοντος από τη Βουλή των Λόρδων. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα κύριε Δεκάστρο για την πρόσκληση που μας απευθύνατε να συζητήσουμε σήμερα αυτό το σημαντικό ε, ζήτημα σε μια κέρια στιγμή και ευχαριστώ και τον Επιτροπό που ήρθε να συζητήσει μαζί μας. Η Επιτροπή μας, η Υποεπιτροπή της Βουλής των Λόρδων για την Γεωργία, δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα μια έκθεση για την καινοτομία στην ε, Γεωργία της Ένωσης. Κάλυψε πολλά ζητήματα, προφανώς και το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, λάβαμε πολλές προτάσεις και θα ήθελα να αναφερθώ σε μία και διαβάζω από μέσα η οποία έλεγε πως εμείς στην Ευρώπη καθόμαστε και λέμε πως η γεωργία είναι η παλιά οικονομία σε αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα ένα εχθρικό περιβάλλον. Πολλές πολιτικές ομάδες μας λένε να πάμε πίσω στον 19ο αιώνα γιατί θα είναι καλό για το περιβάλλον. Αλλά πρόκειται για μια στρατηγική συζήτηση. Λέει η Ευρώπη πως μπορεί να θρέψει 500 εκατομμύρια πλούσιου Ευρωπαίου και να κάνουμε εισαγωγέ ή θα παίξουμε ένα ρόλο στη διατροφή 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων και των Ινδών και των Κινέζων που αρχίζουν να τρώνε κρέας. Οπότε συμφωνούμε πως η καινοτομία πάει πράγματι στην καρδιά της απάντησης η οποία απαιτείται εάν είναι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια ένωση καινοτομία μέχρι το 2020 και ειδικά η πρόταση η οποία κατατέθηκε για μια για μια σχέση καινοτομία. Και ελπίζω ο κύριο Επίτροπο ε, να συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνα για να γίνουν τα λόγια πραγματικότητα. Όσον αφορά την ε, κοινή γεωργική πολιτική, θα πρέπει να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής μειώνοντα το ε, ποσοστό της κοινωτική χρηματοδότησης. Εντός του υπόλοιπου προπολογισμού θα πρέπει να ανακατεμηθούν τα κονδύλια από τον πυλώνα 1 στην, στον πυλώνα 2 για την πολιτική καινοτομία. Η δε υιοθέτηση των ε, υπαρξών τεχνολογιών ε, είναι ελλειπής και ζητάμε περισσότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αγρότες που θα αυξήσουν μακροπρόθεσμα το αγροτικό εισόδημα. Οπότε ελπίζουμε η γεωργία να ανέβει ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κύριε Επίτροπε έχετε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για να γίνει σαφής και σεβαστή η ανάγκη προώθησης της καινοτομίας στην γεωργία και εντός κομισιών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Λόρδο Κάρτερ και τώρα σπεράσουμε στην Γαλλική Γερουσία και με ικανοποίηση θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ε, Οικονομικής Επιτροπής ε, και Φόρου Ανάπτυξης, ε, τον κύριο Ζαμπόλε Μωρή. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, δεν θα σας εκπλήξω λέγοντας ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι για τη Γαλλία και για τη Γερουσία συγκεκριμένα μίσον θέμα. Εμείς ε, προσπαθήσαμε να τοποθετηθούμε ε, απέναντι στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Ε, η ΚΑΠ έχει χάσει πάσα αναγνωσιμότητα και έχει αποδυναμωθεί. Τώρα θα πρέπει την ΚΑΠ να την ε, θεωρήσουμε μια ε, πολιτική για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περήφανη, ε, προσφέρει τρόφιμα στον πληθυσμό και δραστηριοποιείται μέσα σε ένα περιβάλλον που αποτελεί κοινή κληρονομιά. Ε, προτείνουμε να αναδιαρθρωθεί η ΚΑΠ σε δύο, πρώτους, σε δύο κύριους πυλώνες. Ε, καταρχήν ε, να έχουμε μια ασφαλή και ποιοτική γεωργική παραγωγή με κατάλληλο εισόδημα για τους αγρότες ε, και δεύτερον να λάβουμε υπόψη τους περιβαλλοντικούς και τους οδοφυκτικούς παράγοντες. Αυτή η πολιτική μας ε, οδήγησε στο να, εκφράσουμε κάποιες επιφυλάξεις για το πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα. Θέλουμε τα πράγματα να τα βάλουμε στο σωστή του θέση. Αυτή η θέση εκφράζεται σε μια έκφραση που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2010 και που αναφέρεται και στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Τώρα, μετά την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν, τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν ε, την αποστολή να τοποθετηθούν ε, σε σχέση με το θέμα αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι θα είμαστε πιο ισχυροί αν λειτουργήσουμε από κοινού. σήμερα θα πρέπει να δημιουργήσουμε συμμαχίες, το κατάλαβαν οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια θα πρέπει να το κάνουν με τη σειρά τους. Είμαι πολύ περήφανος που το Γαλλικό Κοινοβούλιο και η Γερμανική θα κατέληξαν σε κοινή δήλωση για την ΚΑΠ. Ο, καταρχήν, ο στόχος της επισητιστικής ασφάλειας ε, είναι στρατηγικός. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σύγκληση στα επίπεδα της ενίσχυσης και να δεκτούμε όχι μόνο την εγκατάληξη των ιστορικών αναφορών ή μαζί της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να γίνεται ε, μέσα, μέσω της κατάλληλης ρύθμισης. Ε, αυτή η δήλωση τη πρώτη πολλών δηλώσεων που ελπίζω να ακολουθήσουν. Συνεργαζόμαστε και με το Ισπανικό Κοινοβούλιο και με την Ιταλική Γερουσία και είμαστε και ανοιχτοί στα υπόλοιπα κοινοβούλια. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τώρα ας περάσουμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Ρουμανίας και με ικανοποίηση θα δώσω το λόγο στην ε, Πρόεδρο της Επιτροπής ε, Γεωργίας και Δάσος, Στέλια Φουτζία. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την διοργάνωση αυτής της ε, συνάντησης. Η Κομισιόν έχει πάρα πολύ δύσκολη δουλειά εδώ πέρα για να βρει έναν συμβιβασμό. Ακούστηκαν ήδη πολλές ε, απόψεις και καλό θα είναι να καταλήξουμε σε ένα λογικό συμβιβασμό η Ρουμανία θεωρεί σημαντικό να διατηρηθούν οι δύο πυλώνες με το ύψος ε, που έχουν τώρα από πλευράς κονδυλίων και βέβαια χρειαζόμαστε μια βελτίωση της ε, παραγωγικότητας. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να σκεφτούμε την χρήση βιοτεχνολογιών που ε, ήδη εδώ και πολλά χρόνια αποτελούν αντικείμενο έρευνας η Ρουμανία θα ήθελε οι γεωργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν και στο εσωτερικό της Ένωσης και παγκοσμίως ή ε, συνθήκες ανταγωνισμού. και βεβαίως ε, χρειάζεται στήριξη και η πολιτική και η πολιτική υπερφυριακή και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η σύγκληση μέχρι και πέρα από το 2016 ε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια πολιτική ε, δύο καταγοριών και κάποιοι, να, κάποιοι γεωργοί να βρίσκονται αν θέλετε στην ε, business και κάποιοι άλλοι να κάθονται στην οικονομική θέση. Έχουμε έτσι μια Ευρώπη δύο κατηγοριών ενώ θα έλεγα πως βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο αεροπλάνο θα το τοποθετούσα έτσι. Χρειάζεται επίσης ε, μία μείωση της ε, γραφειοκρατίας και ενίσχυση των εξαγωγών και θα πρέπει να σκεφτούμε πως υπάρχει πέρα από την ευρωπαϊκή και η παγκόσμια αγορά. Λοιπόν, έχουμε ακόμα τρει ομιλητέ και τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Τώρα θα δώσω το λόγο στον στην εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου της Πολωνίας, πρόεδρο της ε, Επιτροπής ε, Γεωργίας, ε, Κορσενιόφσκι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας ε, καλέσατε σε αυτή την ε, ακρόση σήμερα. Και θέλουμε να πούμε ότι η Πολωνία πάντοτε ήταν υπέρ μια ε, ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική με έναν ισχυρό προπολογισμό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η κοινή γεωργική πολιτική αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις γιατί αν αναφέρουμε τα λόγια του κ. Σαβίσκη που τα αναφέρει και ο κ. Δέστ ε, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την κοινή αγροτική πολιτική. Και ε, αυτό φάνηκε και από τις παρεμβάσεις που ακούσαμε σήμερα. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο ομάδες, τα παλιά και τα νέα κρατημέλη οι χώρες έχουν τεράστιες προσδοκίες ε, και ε, οι παλιές χώρες ε, έχουν μια ρεαλιστική συμπεριφορά σε έναν βαθμό που μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό, αλλά σε επανέλθουμε στην έκθεση του κυρίου Ντες και να δούμε ποιο, το, ποιο είναι το πρόβλημα με το πρασίνισμα. Εμείς στην Πολωνία μπορώ να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ σκεπτικοί απέναντι στην εκθεσή σας. Ήδη Έχουμε πάρει το μαθημά μας από τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Η συνάδελφος, από, η συνάδελφος από τη Σουηδία είπε ότι ε, μεταξύ του περιβάλλοντος ε, και της γεωργίας θα πρέπει να υπάρχει στενή σύνδεση όμως εμείς στην Πολωνία έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα γιατί η οικονομία μας βασίζεται στο λιγνίτη και φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουμε παρόμοιο πρόβλημα και με το πρασίνισμα τεράστιο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν παρακαλώ να προσέξετε πάρα πολύ πώς θα επιλύσετε το πρόβλημα γιατί εμείς δεν θέλουμε να υποστούμε τρομακτικές συνέπειες. Παρόμοιες συνέπειες όπως συνέβη με την νομοθεσία της Κομισιόν ε, για το διοξείδιο του άνθρακα για τις σχετικές εκπομπές. Τώρα δεν θέλω να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί και το θέμα της ζάχαρης και του γάλακτος φυσικά. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για ορισμένα κράτη-μέλη και συγκεκριμένα για τη χώρα μου. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, θα δώσουμε τώρα το λόγο στον πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ρούμπιξ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ και δύο χρόνια σχεδόν συζητάμε την ε, κοινή γεωργική πολιτική και τις ε, προοπτικές της μέχρι το 2020. Όλα αυτά συμβαίνουν σε γενικούς όρους. Εντάξει, όσο είναι σε γενικούς όρους δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλοι συμφωνούν ότι θα έπρεπε να έχουμε μέτρα του λεγόμενου πρασινίσματος, να είναι πιο δίκαιη η κατανομή των πληρωμών, αλλά μόλις στάσουμε στην ουσία και στα νούμερα, δεν συμβαίνει το ίδιο. Οπότε αυτά τα οποία ακούσαμε χτες από τον ε, κύριο Επίτροπο. Δεν ε, νομίζω πως ε, είναι θετικά για τους 133.000 ε, γεωργούς στην Λετωνία. Λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή 33% του ύψους των μέσων άμεσων πληρωμών και το 2020 θα λαμβάνουμε 52%. Είναι δίκαιο αυτό έχουμε την καλύτερη καλλιεργήσιμη γη ή μήπως το καλύτερο κλίμα. Αυτό το οποίο λοιπόν θα ήθελα να πω είναι πως ε, όλα αυτά τα οποία ε, υπόθηκαν ε, σε γενικές γραμμές στις τρεις αυτές εκθέσεις είναι πάρα πολύ σωστά και εγώ σέβομαι τους εισηγητές αλλά όταν θα φτάσουμε να γίνουν τα λόγια πράξη θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας περάσουμε στο ε, Βουλή της Αυστρίας και θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Υποτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα σε αντίθεση με τον συνάδελφο από τη Γερμανία. θεωρώ πως ε, το πλαφόν είναι βασικό μέτρο για την δικαιοσύνη. Γιατί ξέρετε πως ε, αλλιώς δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος γιατί θα πρέπει να οδηγηθούμε στο μέλλον προς οποιαδήποτε γεωργία και του πρασινίσματος και οτιδήποτε άλλο. Εάν δούμε λοιπόν την έκθεση Lion, την έκθεση DES και το έγγραφο των επιλογών, βλέπουμε πως υπάρχουν ε, πάρα πολλέ δηλώσει για προστασία του κλίματος, περιβάλλον, βιοπικιλότητα, αλλά κυρίε και κύριοι έχουν όνομα όλα αυτά και λέγονται βιολογική γεωργία. Ο παλαιός κανονισμός 834 αποτελεί θεμέλιο νομίζω για τη γεωργία του 21ου αιώνα. Πού είναι η φιλόδοξη προσέγγιση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία μόνο φορά σε μία παρένθεση στην έκθεση DES αναφέρεται η λέξη οικολογική γεωργία. Όχι, δεν αρκεί αυτό, είναι πάρα πολύ λίγο. Και κατόπιν ε, προς τον Βρετανό και τον Ρουμάνο συνάδελφο. Μία γεωργία χωρίς γενετικά τροπημένους οργανισμούς είναι αυτό το οποίο θέλουν οι πολίτες ε, και οι καταναλωτές. Δεν υπάρχει πρασίνισμα με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν είναι λύση αυτή για το μέλλον. Και το έχουν αναγνωρίσει πολλά κράτη-μέλη, πολλές περιφέρειες και χαίρομαι ήδη για το ότι ο Επίτροπος ο κ. Τσόλος ξέρει πως δεν είναι αυτός ο δρόμος της ποιότητας. Είναι σημαντικό και πρέπει να εμβαθύνουμε άρα συμπεριτέρω συζήτηση σε αυτό το πλαίσιο. Και τέλος μία λέξη για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Κοιτάξτε, όλοι ως εκπρόσωποι της Γεωργίας στα κοινοβούλια μας ε, έχουμε μια σημαντική ε, αποστολή. Να φέρουμε την Κομισιόν σε αυτό το οποίο είναι σημαντικό για εμάς, τον φόρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Και εκεί πέρα θα βρεθούν τα λεφτά και πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό. Και δεύτερον, περισσότερα λεφτά για την γεωργία. Να φύγει αυτό το συνολικό πλαφόν στο γεωργικό προϋπολογισμό, να έχουμε περισσότερα χρήματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, θα επανέλθουμε στη Γερμανία. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Όλικ Χόφιλ που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τη Γεωργία και την Πολιτική των Καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως Γερμανίδα θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα. Η γεωργική πολιτική έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία και από πλευράς ε, Ασφάλεια των τροφίμων αλλά και για να έχουμε μια αηφόρο ασφάλεια των ε, τροφίμων και βεβαίως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις σπατάλη των ε, τροφίμων και να σταματήσουν βεβαίως και οι απώλειες και να μην ε, ρίχνουμε και μεγάλες μάζες στις παγκόσμιες αγορές αλλά βεβαίως συζητάμε και το πρασίνισμα το τι περιέχεται στην ε, πρόταση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεχόμαστε. Μιλάμε επίσης για την απλοποίηση. Νομίζω πως ε, μπορούμε να μιλήσουμε και μια στρατηγική πρωτεϊνών που μπορεί να συνδεθεί με το πρασίνισμα αυτό, αλλά σημαντικός είναι και ο δεύτερος πυλώνας, το ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα τα οποία περιέχουν πολλά καινοτόμα μέσα όπως παραδείγματο χάρη ενεργειακές υπηρεσίες αλλά και ο περιφερειακός χαρακτήρας, στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δεν μπορούν να ή δεν θέλουν να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Αυτό σχετίζεται με τον δεύτερο ε, πυλώνα που δυστυχώς εδώ πέρα δεν υπάρχει στο ψήφισμα. Η δε διάσκεψη των ε, Γερμανών ε, Υπουργών Περιβάλλοντος. Κοιτάξτε, είναι διαφορετική κατάσταση στη Γερμανία. Στην ε, Ρινανία, Παλατινά, το από όπου προέρχομαι, το θεωρούν κάτι το σωστό το πλαφόν και θεωρούν πως θα υπάρξει και δικαιοσύνη εντός της Γερμανίας. Τώρα όσον αφορά τους κανονισμούς ε, αγοράς ε, θέλω να συμφωνήσω με εκείνους που βλέπουν επικριτικά την απορρίθμιση. Συζητάμε και για την ζάχαρη, δηλαδή για την παράταση για τον ε, ίνο επίσης, αλλά και για το γάλα. Θα πρέπει εδώ πέρα να επανεξετάσουμε τα πράγματα και πιθανώς να πάμε σε μια νέα κατεύθυνση. Όσον αφορά την έρευνα, πρέπει πράγματι να αυξηθεί η σημασία της έρευνας, αλλά όχι η γενετική τεχνολογία, όπως υπάρχει και στη Γερμανία, αλλά καινοτόμα μέτρα στο πλαίσιο της αηφορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα, θα κάνουμε 10 λεπτά διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο γύρο της συζήτησης. Ευχαριστώ όλους. <laughs> It's not easy to manage, but uh, uh, uh I need you. Yeah.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 Allora riprendiamo i lavori e molto Μπορούμε να ξαναρχίσουμε και θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους ε, του Κυπριακού Κοινοβουλίου, πρόεδρο της ε, Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, τον κύριο Γιαννάκη Γαβρίλη. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Επιτρέψτε μου να εκφράσω τι θερμέ μου ευχαριστίε προ την Επιτροπή Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρωτοβουλία τη διοργάνωση τη σημερινή συνάντηση. Η μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική είναι επίκαιρο και κρίσιμο θέμα που μα απασχολεί και μα προβληματίζει όλου. Η Κύπρο υποστηρίζει τη δικαιότερη κατανομή των δημοσιονομικών πόρων στα κράτη-μέλη στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα λαμβάνουν υπόψη τι επιπτώσει της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη με απότερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι η διασφάλιση της παροχής στοχευμένων επιδοτήσεων. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει επίση να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα τη κοινοτική γεωργία με την παροχή κινήτρων που αποσκοπούν στην ευθάριση των νέων να ασχοληθούν με το επάγγελμα του γεωργού και τα άλλα ταμεία μέσα από τη λήψη μέτρων κοινωνική συνοχή τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση στην Ήπεθρο μπορούν να συνδράμουν καταλητικά προ την κατεύθυνση τη ευθάριση των νέων να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Οι άμεσε πληρωμέ θα πρέπει να κατανέμονται στη βάση πιο δίκαιων κριτηρίων, οι οποίε έχουν ήδη αρνητικό αντίκτυπο στην Κύπρο, όπω και αλλού. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στι εκμεταλλεύσει τη υπαίθρου, εφαρμόζοντα ανώτατο όριο στήριξης ανακμετάλλευση. Οι διαδικασίε θα πρέπει να απλοποιηθούν και να είναι ευέλικτε, με τρόπο που να επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να προσαρμόζουν την πολιτική των άμεσων πληρωμών στι ιδιαιτερότητε του. Ομολογουμένω, η γεωργία δεν είναι απλώ ένα τομέα παραγωγή που επηρεάζει αποκλειστικά την οικονομική επιβίωση μια ομάδα ανθρώπων, αλλά μια πολυσύνθετη δραστηριότητα που έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο ω αποτέλεσμα του πολυλειτουργικού τη χαρακτήρα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Και τώρα είναι η σειρά του Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Έστερ Τίξο από την Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για τη διοργάνωση της ε, σημερινής σύσκεψης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Υπουργό για τις αρχικές παρουσιάσεις τους. Η Εστονία πιστεύει πως ε, η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει μια πραγματικά κοινή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίδια για όλους. Επίσης, ε, θα πρέπει να καταστήσουμε δικαιότερες ε, τις άμεσες πληρωμές, διότι μέχρι στιγμής παρατηρούνται πολύ σοβαρές ε, διαφορές ε, και αυτό στρεβλώνει την ε, εσωτερική αγορά. Κατά την μεταρρύθμιση της πολιτικής θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στον παραγωγό, στο ρόλο που διαδραματίζει στην αλυσίδα εφοδιασμού. θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί η ίδια η βάση της γεωργικής πολιτικής ε, και να επενεξεταστούν οι δύο πυλώνες. Με τα τελευταία νέα δε, τα χθεσινά νέα για τον ε, προϋπολογισμό, δυσκολεύει η κατάσταση. Η νέα μεταβατική περίοδος ε, δε είναι επιζήμια για τους γεωργούς μας. Υποστηρίζουμε επίσης την έρευνα και την καινοτομία για το ρόλο που έχουν στην γεωργική πολιτική. Από την Ιταλική Γερουσία τώρα, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, ο Γερουσιαστής Αλφόνσο Άντρε. Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφοι, θέλω να εκφράσω την εκτίμηση μου για την πρωτοβουλία του Πρόεδρου Δικάστρο και τη Επιτροπή του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο που προσπαθήσαν ε, να ε, προβούν σε, μια, σε ένα διευρυμένο προβληματισμό για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η ε, μεταρρύθμιση της ΒΕΚ, η Γερουσία της ε, Ιταλικής Δημοκρατίας ε, συνεισφέρει με την ε, εκπόνηση μιας συμπεφωνημένης εθνικής θέσης και μαζί με τον συνάδελφο Ρεσο Πιντζόνα προσπαθήσαμε να συγκλίνουμε για ορισμένα θέματα ιδιαίτερα σημαντικά. Θα πρέπει η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να επικεντρωθεί στα μέτρα της αγοράς, της άμεσης ενισχύσης και στους άξονες της αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με μια νέα διάφρωση που να στοχεύει στην εφαρμογή των διεκασιών και στο να τεθεί τέλος ε, των αμέσων ισχύσεων για τους επαγγελματίες γεωργούς ε, υπέρ της δημιουργίας θέσεων εργασίας ε, και υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Πρέπει να αντιμετωπίσει η γεωργία τις παγκόσμιας προκλήσεις και θα πρέπει να στραφεί στην έρευνα και στην κοινοτομία να υποστηρίξει την απασχολησιμότητα των γυναικών και των νέων. Εγώ θα έλεγα να μην, να μην ξεχάσουμε το θέμα της εργασίας και να θεωρήσουμε ότι είναι κύριο το ζήτημα αυτών των θέσεων απασχόληση. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά σχετικά στοιχεία στην ανακοίνωση ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρουσιάστηκε από τον Επίτροπο Τσόλο τον Νοέμβριο του 2010. Όμω χρειάζεται πρόσθετη προσπάθεια. Η ορθή οδό είναι αυτή που διανύουμε σήμερα και να εξαλείψουμε την αναποτελεσματικότητα και την ανισότητα και έτσι ώστε η ΚΑΠ να γίνει μια πραγματική πολιτική πρόθεση του δημοσίου αγαθού σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σεστιάντρια και τώρα θα περάσουμε στους εκπροσώπους του Ολλανδικού Κοινοβουλίου και θα δώσω το λόγο στον κύριο Έρικ Σμάλινγκ. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και διδακτικά αυτά τα οποία ακούσαμε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ντες ε, για το έργο του και είναι καλό να γνωρίζουμε πως βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις για τον πρώτο πυλώνα και τις ανησυχίες των ε, συναδέλφων από την Ανατολική Ευρώπη. Η Ολλανδία είναι ιδρυτικό μέλος, όπως ξέρετε, της ένωση Έχει επωφεληθεί πάρα πολύ από την κοινή αγροτική πολιτική και πραγματικά θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρξει εδώ πέρα πολύ περισσότερη αλληλεγγύη. Είναι καλό δηλαδή το επίπεδο της φιλοδοξίας που υπάρχει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει νομίζω και μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα, θα ήθελα να πω πως α, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος κίνδυνος γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει πως δίνει σε εθνικό επίπεδο αυτά τα λεφτά σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα π.χ. θα μπορούσε να είναι τα αμμόδια εδάφη που έχουμε στην Ολλανδία, κίνδυνος πλημμύρες ε, και άλλα χαρακτηριστικά ολλανδικά. Οπότε θα ήθελα να ε, αναζητήσουμε κάποιους κοινούς στόχους όσον αφορά τον ε, δεύτερο πυλώνα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο είπατε για την πράσινη Φιλανδία και τη λιγότερο πράσινη ε, Σικελή, αλλά νομίζω πως μπορεί να βρεθεί κάποιο κοινό εδαφός κατόπιν. Να αναφερθώ στην ε, σύνδεση του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου και αυτών των οποίων είπε ο κύριος Πίμπαλ. Σα ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο τώρα σε πρόσωπο ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Δανέλη. Ε, αγαπητέ Επίτροπε, που δεν είναι εδώ, αγαπητέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω δύο σύντομε παρατηρήσει: Οι προτάσει τη Επιτροπή για τον προπολογισμό τη κοινη γεωργικη πολιτική πολιτικής 14-20 ε, φυσικά και δεν εγγυώνται την τελική μορφή που αυτές θα πάρουν. Ούτε όμως βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ε, προβλέπεται να ε, εφαρμοστούν πολλές από αυτές τις ε, νέες προβλέψεις και προτάσεις. Όμως οφείλουμε να ενθαρρύνουμε και να στηρίξουμε τις κατευθύνσεις αυτών των προτάσεων γιατί νομίζω ότι πολλές από αυτές είναι φανερό ότι αέρουν στρεβλώσεις ή ανεπάρκειες της σημερινής κοινή γεωργικής πολιτικής. Και δεύτερο, νομίζω και είναι θετικό να το επισημαίνουμε ότι όλο και περισσότεροι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιλαμβάνονται ότι το πραγματικό δίχτυ ασφαλείας δεν έχει να κάνει μονάχα με τις άμεσες ενισχύσεις, αλλά κυρίως ζητούν από μας μέτρα στήριξης των προ... εκείνων ώστε να παράγουν ποιοτικά, επώνυμα και ανταγωνιστικά προϊόντα που να μπορούν να βγουν σε μια δύσκολη και όλο και περισσότερο απαιτητική αγορά μέτρα στήριξης ώστε να μπορούν οι ίδιοι να καρποθούν όσο γίνεται περισσότερο της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων τους. Ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστώ Σπύρο. Να περάσουμε τώρα στη Γερμανική Bundestag και θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Φρίντρικ Ωστεντολφ. Ja, ε, Ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές στη Γερμανία δεν έχουν όλοι μία άποψη για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει μεταρρύθμιση. Έχουμε την πρόκληση ε, του Επιτρόπου Τσιόλος και χαιρόμαστε για το ότι είναι στο πλευρό μας. Ε, πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά τη γεωρική πολιτική. Επίσης θεωρούμε πως εμείς ως παράσινοι είμαστε ε, υπέρ του να ενισχυθούν τα ερωτήματα που, και τα ζητήματα που θέτει η κοινωνία στους αγρότες για να συνεχίσει να πληρώνει την γεωργία. Και βεβαίως σε αυτό ανήκει και η προστασία των ζώων που θα παίξει σημαντικό ρόλο, ήδη παίζει μεγάλο ρόλο στη Γερμανία στο μέλλον για να συνεχίσει να υπάρχει αποδοχή της ε, γεωργίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει Βλέπετε πως υπάρχουν ορισμένες φορές σε κάποια χωριά σχεδόν πολεμικές αντιπαραθέσεις ε, όταν υπάρχουν μεγάλες μαζικές εγκαταστάσεις ε, κτηνοτροφικές. Αυτό ε, για τη συζήτηση. Πράγματι πρέπει να το δούμε αυτό στη μεταρρύθμιση, αλλά υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της βιοπικιλότητας, το οποίο εξακολουθεί κατά την άποψή μας να μας απασχολεί. Εντάξει, η κλιματική αλλαγή ε, μεγάλη πρόκληση, αλλά εξίσου μεγάλη είναι και η βιοπικιλότητα. Η βιοπικιλότητα δημιούργησε η γεωργία, αλλά την καταστρέφει κιόλα ταυτόχρονα. Και αυτό πρέπει να το δούμε σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια και με περισσότερες αποχρώσεις. Οπότε για εμάς, ε, ειδικά στον πρώτο πυλώνα, το πρασίνισμα είναι ζήτημα υπαρξιακό. Γιατί εμείς ε, στη Γερμανία συζητάμε εσωτερικά μήπως το έπρεπε θα προχωρήσουμε σε ακόμη μεγαλύτερες ε, μειώσεις ε, και πέρα από ένα 70%. Τώρα μια τελευταία παρατήρηση για το πλαφόν στις ε, πληρωμές. Εμείς θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνει. Βεβαίως παλεύουμε μια συμμαχία σοσιαλδημοκρατών, κομμουνιστών και δεξιών σε μια σπάνια συμμαχία. Ε, εμείς και οι φιλελεύθεροι είμαστε κατά, ε, υπέρ με συγχωρείτε, του πλαφών. Δεν είναι δυνατόν 1500 ε, εκτάρια να παίρνουν 450.000 ευρώ και να δουλεύουν σε αυτά 5 άτομα ενώ σε μια άλλη χώρα να παίρνουν 12.000 ευρώ. Δεν είναι. Δικαιολογείται αυτό. Bene, grazie. Ευχαριστούμε και ας επιστρέψουμε στην Ελλάδα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χατζόσμαν, παρακαλώ. Πρόεδρε, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που παραβρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας σε μια εξαιρετικά σημαντική συνεδρίαση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού με τα Εθνικά Κοινοβούλια με θέμα το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον καπνό και συγκεκριμένα για τον μπασμά αυτό είναι και ο λόγο που με φέρνει στην Επιτροπή. Ο μπασμά που καλλιεργείται στην περιοχή μου την Ροδόπη είναι μια παραδοσιακή καλλιέργεια εξαιρετική ποιότητα με αυξημένη ζήτηση στι διετή αγορέ. Περισσότερε από 15.000 οικογένειε απασχολούνται στην μονοκαλλιέργεια του καπνού στην ευρύτερη περιοχή τη τράκη. Οι κλήροι που διαθέτουν είναι μικρή έκταση συνήθω, δεν ξεπερνούν τα 5-10 στρέμματα και οι συνθήκε δεν ευνοούν τη συστροφή σε άλλε εναλλακτικέ καλλιέργειε με τόσα λίγα στέματα. Με τον πασμά ασχολούνται όλα τα μέλη μια οικογένεια, Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια απαξίωση του καπνού. Οι χαμηλέ τιμέ, η αύξηση του κόστου παραγωγή αποτελούν συνεχείς προκλήσει για του παραγωγού μα. Κάτω από αυτέ τι αντίξωε συνθήκε, οι ευρωπαϊκέ επιδοτήσει αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα στο πενικλό εισόδημα των καπνοπαραγωγών και συγχρόνως οικονομική ανακούφιση και αποκούμπη για χιλιάδες ενεργούς παραγωγούς στην περιοχή μου. Η στήριξη του καπνού δεν αφορά μόνο την ενίσχυση 15.000 οικογενειών της Τράκης, αφορά την οικονομία της περιοχής μου, αφορά την οικονομία της Ελλάδας. Στην Τράκη ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον συλλοβάτη της οικονομίας πρέπει να γίνουν οργανωμένες προσπάθειες στηρίξης και ενίσχυσης της γεωργίας. Οι καπνοπαραγωγοί μας σήμερα βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση και έχουν φτάσει στα όρια της φτώχεια και της πείνας. Εκφράζουν έντονα την ανησυχία τους για το μέλλον του Μπασμά, για το μέλλον των οικογενειών τους. Σας καλώ όλους να ε, σκεφτείτε τα όσα υπόθηκαν σήμερα για τον καπνό. Σας καλώ να στηρίξετε το δίκαιο και λογικό αίτημα των παραγωγών για συνέχιση των επιδοτήσεων υπό το καθεστώς της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Λούλινγκ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρεσβύτερη μας εδώ στο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να σας, μιλήσω συγγνώμη, για δύο προβλήματα που θα μας απασχολήσουν και μετά το 2014. Πρώτον, κατάργηση των γαλακτοκομικών ε, πιστο... Ε, ποσοστώσεων. Θα επέλθει η κατάργηση αυτή, αλλά στο ενδιάμεσο μας υποσχέθηκαν ομαλή προσγείωση. Γνωρίζω ότι τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη δεν είναι να εξαντλούν πλέον τις γαλακτοκομικές τους ποσοστώσεις, καθότι η παραγωγή τους είναι χαμηλότερη από τις ποσοστώσεις που δικαιούνται και ακόμη και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παραγωγή είναι χαμηλότερα των ποσοστώσεων. Όμως, σε κάποιες χώρες υπερβαίνει η παραγωγή της ποσοστώσης ε, κατά πολύ και τι σημαίνει αυτό, ότι οι παραγωγοί μας πρέπει να ε, πληρώνουν διαρκώς την συνεισφορά λόγω υπερπαραγωγής ακολουθούσε ευθύνουσα απορία ε, αυτό το τέλος ως συνοδευτικό μέτρο για την κατάργηση δηλαδή των ποσοστώσεων και πιστεύω ότι θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποστηρίξει για αυτήν την ομαλή προσγείωση. Ε, σχετικά τώρα με την κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης μετά το 2015 και το 2018 αντίστοιχα, πράγμα που αντιστοιχεί την ειδική ομάδα του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Στο Στρασβούργο κάναμε διαβούλευση ε, με τους ε, καλλιεργητές, καλλιεργητές ε, οι οποίοι μας είπαν ότι με την κατάργηση των δικαιωμάτων ε, μπορεί να μην επιβιώσουν οι εκμεταλλεύσεις τους, ε, κυρίως οι εκμεταλλεύσεις που παράγουν σταφίδες ή κρασί καλής ποιότητας στις πλαγιές σε σχέση με το κρασί χαμηλότερης ποιότητας της πεδιάδας με την διεπαγγελματική αναδιοργάνωση των ε, ίνων της ε, Καμπανίας. Α, και να σας πω ότι η Σάντι ε, δημοσίευσε ένα πολύ μνησί κακό άρθρο με διάφορες ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις. Έχω γίνει στάρ στο Βρετανικό τύπο πια. Ε, τι πρέπει να κάνει κανείς για να είναι γνωστός στο πολιτικό στερέωμα. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τη θέση μου. Σας λέω πάντως ότι στην Καμπανία, στην περιοχή της Καμπανίας, τέσσερις ώρες ε, μας βομβάρδιζαν σε ένα σεμινάριο. Ε, τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες τώρα για την ποιότητα του σεμιναρίου, αλλά πάντως ακούσαμε τους φόβους και τις ανησυχίες των αμπελουργών για, αυτή τη δυστυχή ατυχή λύση στην οποία κατέληξαν οι Υπουργοί το 2008 διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν κατά μεν τότε, αλλά δεν είχε το δικαίωμα συναπόφαση ε, δε. Ήταν μια άθλια συμβιβαστική λύση ε, του Συμβουλίου για τα δικαιώματα φύτευσης ε, και ήταν άθλια για όλες τις περιοχές. Ε, πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτή τη θέση το ταχύτερο δυνατόν. Ο Επίτροπος όλος απο, αποχώρησε δυστυχώς, αλλά ίσως συνεργάτες του μπορούν να το διαβιβάσουν το μήνυμα, γιατί όπως λέμε και στην έκθεση του κυρίου Ντες και τον ευχαριστώ. Θέλουμε στο πλαίσιο των ε, νομοθετικών προτάσεων που αναμένουμε για το φθινόπωρο να συμπεριλάβει πρόταση για κατάργηση αυτού του συστήματος, αλλιώς θα υποβάλουμε τροπολογίες και θα υπεραμεθούμε τις θέσεις μας, σας διαβεβαιώ, για τον προϋπολογισμό τώρα. Ε, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Ένα θα τονίσω μόνο. Η, δεν είναι η κοινή γεωργική πολιτική που κοστίζει. Η απουσία της, η απουσία της ε, θα επιφέρει ένα ε, δυσβάσταχτο άχθος για την κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική Ευρώπη. Το λέω απευθυνόμενο στο συνάδελφο τον Αυστριακό η εισαγωγή νομίζω φόρου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα αποτελέσει τη διάσωση της κοινή ε, αγροτικής πολιτικής. Και βεβαίως ε, δεν ξέρω εάν θα ε, το καταφέρουμε αυτό, φοβάμαι πως δεν είναι Ευχαριστώ κύριε Λούλινγκ. Εσείς μπορείτε να μιλάτε όσο θέλετε, μας εκπροσωπείτε όλους άλλωστε. Λοιπόν, και τώρα θα ολοκληρώσουμε δίνοντας το λόγο στους εκπροσώπους του Εθνικού Κοινοβουλίου της Γαλλίας, τον αντιπρόσωπο ε, της Επιτροπής για τις Οικονομικές Υποθέσεις, τον κύριο Ζαν Γκουμπέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι συνάδελφοί μου από ε, τα γαλλικά κοινοβούλια ε, εξέφρασαν τη θέση της Γαλλίας, αλλά θα περιοριστώ σε δύο ε, θέματα. Σε σχέση με το σχέδιο του Επιτρόπου όλους ε, άκουσα εδώ από τους συναδέλφους ότι ζητούσαν τη σύγκληση, έχουν δίκιο. Ε, θα πρέπει να εγκρίνουμε το πρασίνισμα και είναι και λογικό να δώσουμε και περαιτέρω μέσα και εργαλεία στην έρευνα, όμως όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα περιορισμένο προϋπολογισμό και κάποια στιγμή αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες θυσίες. Και αυτή είναι η θέση της Γαλλίας. Εγώ νομίζω ότι, ε, ότι, ε, ότι τελικά θα υπάρχουν σημεία σταδιακής, μέτρα σταδιακής μείωσης, γιατί αν το κάνουμε τελικά οι αγρότες των πιο μικρών χωρών θα πληρώσουν πιο ακριβά τη μεταρρύθμιση. Έτσι λοιπόν ε, το πακέτο αυτό δεν ε, είναι αναγκαστικά να το δεκτούμε ή να το αφήσουμε, αλλά ε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε το συνολικό πνεύμα αυτού του πακέτου. Τώρα δεύτερη παρατήρηση αφορά κάτι διαφορετικό. Δεν αφορά τόσο την σημερινή συζήτηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πω. Εμεί ζητάμε από του ε, αγρότε μα να σέβονται διάφορου ε, κανόνε για την παραγωγή, για την προστασία του περιβάλλοντο, ε, ηθικού κανόνε κτλ. Όμω πολλοί από αυτού, δεν καταλαβαίνουν πώ δεν έχουμε τι ίδιε απαιτήσει για τα προϊόντα που εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα που έρχονται από τι άλλε περιοχέ του κόσμου δεν σέβονται του ίδιου κανόνε. Και Πιστεύω, αν δεν έχουμε αυτό τον παραλληλισμό ε, τύπης, όπως λέμε ε, στη Γαλλία, νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη παρανόηση και παρεξήγηση από την πλευρά των γεωργών, αλλά και των καταναλωτών που θα καταλαβαίνουν ότι δεν ε, προστατεύονται τόσο καλά από την Ευρώπη όπως θα έπρεπε. Σας ευχαριστώ. Συμφωνούμε απόλυτα για το θέμα αυτό. Είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση του κ. Παπαστάμκου που Ουσιαστικά δέσμευε τα ευρωπαϊκά όργανα να σέβονται τους κανόνες της αμοιβαιότητας. Οι δικοί μας γεωργοί σέβονται πάρα πολύ ψηλά πρότυπα, αλλά ε, πρέπει να δούμε το αν υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός με τις αγωγές από άλλες χώρες, γιατί οι υπόλοιποι δεν σέβονται τέτοια πρότυπα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Εθνικού Κοινοβουλίου, πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας, τον κύριο Σάντορ Φόντ, για δύο λεπτά. Köszönöm szépen, köszöntöm a szervezőket του, Κοινοβουλίου θα ήθελα να σα χαιρετήσω όλου. Ε, συμφωνούμε με τι ε, βασικές αρχέ ε, τη μελλοντική μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε να επαναληφθούν λάθη του παρελθόντο. Γιατί δεν μπορούμε να δυσκολεύουμε τη ζωή των αγροτών και των κτηνοτρόφων έτσι ώστε τελικά να εγκαταλείψουν ε, τη γεωργία. Και αυτή η έννοια του παρσινίσματος, ε, του greening, ε, αν είναι υπερβολικά αυστηρή θα μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες συνέπειες. Έγινε λόγο και για τον αμπελονικό τομέα προηγουμένω. Ε, εισάγονται προϊόντα από τέτοιε χώρε ε, που παραγόνται υπό ε, συνθήκε που είναι άγνωστες εμάς ή παραδείγματο χάρη μπορεί να έχουμε άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε του αγρότε και τους κτηνοτρόφους και πρέπει τα προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες να σέβονται τους ίδιους κανόνες που ισχύουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχουν ε, λάβει η χώρα λάθη, έχουν γίνει λάθη στις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη τα δικαιώματα φύτευσης και την απελευθέρωση του ελληνικού τομέα. Η Ουγγαρία δεν συμφωνούσε. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τη μεταρρυθμίση για τα ζαχαρότευτλα. Κάθε φορά γίνεται πιο δύσκολη η ζωή των αγροτών και των κτηνοτρόφων γιατί οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις διανομής είναι αυτές που τελικά ελέγχουν ε, τις τιμές της αλυσίδας και αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Έτσι λοιπόν ζητούμε από όλου, από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Κομισιό, να μην δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα στους γεωργού και στους κτηνοτρόφου από όσα ήδη αντιμετωπίζουν. Δεν ε, μπορούμε να παρουσιάζουμε και να θέτουμε περισσότερες δυσκολίες στους ανθρώπους αυτούς. Οι ε, νέοι γεωργοί ε, Ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα όπως η σημερινή γενιά, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να ασχοληθούν με τη γεωργία. Θα πρέπει να δώσουμε ε, τις δυνατότητες αυτές στους ανθρώπους και επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε την επιστηστική ασφάλεια για όλους τους Ευρωπαίους. Μάλιστα, τελειώσαμε το γύρο ε, των παρεμβάσεων ε, έχουμε ορισμένους εκπροσώπους από το Εθνικό Κοινοβούλιο που ζητούν να ξαναπάρουν το λόγο. Υπάρχει τέτοια βούληση. Διαφορετικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώνεται εδώ αυτή η σημαντική σημερινή συνεδρίαση που μας επέτρεψε να γνωρίσουμε καλύτερα τις ευαισθησίες ε, όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θέλετε και πάλι το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Από την Αυστρία, αντιπρόεδρο της Επιτροπή Γεωργίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα για την Γαλλίδα συνάδελφο που αναφέρθηκε στον φόρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Κοιτάξτε, και εγώ υποθέτω πως θα πρέπει να προωθηθεί με δικά της μέσα η κοινή γεωργική πολιτική, αλλά είναι μια σημαντική παρέμβαση στην οποία συμφωνούμε με άλλα κράτη, γιατί όλα τα κόμματα στην Αυστρία συμφωνούν με αυτό το μέτρο. Ήθελα απλά να το ξεκαθαρίσω και να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φόντα από την Ουγγαρία. Η κυριαρχία ή η ασφάλεια των τροφίμων βεβαίως πρέπει να αποτελέσει βασικό σημείο και υπάρχουν πάρα πολλοί δύο θετικά σημεία στην έκθεση Σημείο 8. Εξωτερική προστασία από την ε, ποιότητα. Ναι, εντάξει, αλλά πώς ε, συμβιβάζεται αυτό με τις υποχρεώσεις των ΠΟΕ και ε, στον συνάδελφο Όσντορφ από τη Γερμανία να συμφωνήσω μαζί του και να πω ναι, αυτή οι, αυτές οι φθήνουσες μειώσεις ε, στο σημείο 25 της έκθεσης DES ε, όπως ε, προτείνονται αντικειμενικά είναι μια καλή πρόταση γιατί όλοι γνωρίζουμε πως είναι δεδομένη η αποτελεσματικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων και βεβαίως εκεί πέρα που αναφέρονται οι θέσεις εργασίας και οι αηφόρες διαδικασίες. Νομίζω είναι ένα μοντέλο ε, το οποίο μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την ε, Κομισιόν για να δει παραδείγματο χάρη για τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, βρίσκονται στον μέσο όρο από εκεί και πάνω να υπάρξει μία φθήνουσα να υπάρχει αυτός ο φθήνων χαρακτήρας. Και τέλος όσον αφορά την αποτελεσματικότητα με, την επιπρόσθετα μέτρα, με επιπρόσθετα μέτρα ε, οικολογικά. Θα πρέπει να δούμε βεβαίω και την ποικιλία των καρπών. Και εδώ πέρα νομίζω έχει καλή προσέγγιση η έκθεση. ευχαριστώ. Ωραία. Αν ε, δεν ζητά κάποιο άλλο το λόγο σε σχέση με όσου ήδη παρενέβησαν, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του Πολωνικού Κοινοβουλίου και να του ξαναδώσω το λόγο Πρόκειται για τον ε, γερουσιαστή Γέρση Προσκέψη που θέλει να κάνει μια ανακοίνωση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου ξαναδίνετε τον λόγο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω γιατί εκτιμώ όλος ιδιαίτερο την ευκαιρία που μας δίνεται να ακούσουμε τις απόψεις σας και να είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι για τις εξελίξεις. Τώρα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο μπορούμε να εκπονήσουμε μια καλύτερη νομοθετική πρόταση που να καλύπτει τις ανησυχίες και τις επιθυμίες ε, όλων. Γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω στις 25 και 26 μια συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια όπως αυτή που κάναμε στη Βουδαπέστη για την κοινή γεωργική πολιτική, την επιστημιστική ασφάλεια, για ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλες ε, τις πιθανές ε, λύσεις. Έχουμε ήδη στείλει κάποιες ε, προσκλήσεις στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου θα λάβει η χώρα ε, η συνεδρία σε αυτή και ίσως θα θέλατε να έρθετε κι εσείς για να συμμετάσχετε στη συζήτηση. Μάλιστα, ευχαριστώ. Μου με ενημέρωσαν ότι ήρθε στην αίθουσα και πρόσωπο ε, Κοινοβουλίο από την Βουλγαρία μέλος της Επιτροπής Γεωργίας ε, και Δασών, ε, ο κύριος ε, Πένκο Αθανασόφ. Και του δίνω το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ. Благодаря, господин председател. Няколко думички. Вече явно сме изморени, но... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μόνο κάποιες παρατηρήσεις, ε, λίγες, ε, διότι είσαστε όλοι κουρασμένοι. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε δύο σημεία. Όπως είπε ο Έλληνας ε, συνάδελφος για τον καπνό, ουσιαστικά πρέπει να ασχοληθούμε με ειδικά ζητήματα. Μα όλοι συμφωνούμε για τα γενικά ζητήματα. Όταν όμως περνάμε στα επιμέρους, θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτά που είπε ο Έλληνας ε, συναδελφός για τους καπνοκαλλιεργητές. Ε, στην ε, Βουλγαρία είναι παρεμφερής η κατάσταση για την καλλιέργεια άλλων ανατολικών ποικιλιών καπνού. Οπότε θα ήθελα να το έχετε κατά νου, ανεξαρτήτως απόψεων περί καπνίσματος, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε ότι δεν έχει μειωθεί το κάπνισμα ε, τελικά, τουλάχιστον όχι στην Ευρώπη. Πρέπει να το λάβετε υπόψη. Επίσης ο πυλώνας των άμεσων πληρωμών, ο πρώτος πυλώνας, ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθεί ε, να ληφθούν υπόψη οι διαφορές του παραγωγικού κόστος ανακαλλιέργεια. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η πάπρικα ανά εκτάριο παραδείγμα. Η πιπεριά ανά εκτάριο. 600 ε, ευρώ θέλουμε για την ε, παραγωγή. Ενώ 6 ευρώ μόνο, 60 ευρώ χρειάζονται μόνο για το στάρι. Νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτέ οι διαφορέ. Bene. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώνεται εδώ αυτή η συνεδρίαση που ήταν πάρα πολύ σημαντική συμμετείχαν ε, και 27 Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Εμείς καλούμαστε ναι, όχι μόνο τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων Γεωργών, τα 10 εκατομμύρια, αλλά ε, ε, μιλάμε και για μια απάντηση που πρέπει να δώσουμε σε 550 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ε, εδώ ακριβώς απ' έξω από την αίθουσα έχουμε οργανώσει μια μικρή δεξίωση.